Καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον ε, καθηγητή Ρωμάνο Πρόντι, πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, πρωθυπουργό της Ιταλίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είχε δεχτεί την πρόσκλησή μας για να συνεισφέρει τη συζήτηση που κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την επιστημιστική ασφάλεια. Μία ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρόκληση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της σημερινής ε, συνεδρίασης. Αφορά όλους μας, διότι πρόκειται για μία πρόκληση που αφορά τον κόσμο της γεωργίας, αλλά και τον κόσμο όλης της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινότητας. Στις εργασίες της Επιτροπής αυτής έχουμε συζητήσει επανειλημμένω το θέμα αυτό. Ακόμα και η συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη του το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας. Και σήμερα, αγαπητοί καθηγητή θα συζητήσουμε την έκθεση DES και θα ψηφίσουμε την έκθεση DES που είναι η δεύτερη έκθεση που ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον αυτή της τόσο σημαντικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Στο ψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2010 επαναλάβαμε την δέσμευσή μας για μια ισχυρή γεωργική πολιτική που θα μπορεί να ε, συνεισφέρει στην προάσπιση των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και να έχουμε καινοτομίε και δυνατότητες ε, στο χώρο της υπαίθρου με τη συνεισφορά της ε, γεωργίας για τις άλλε μεγάλες προκλήσεις όπως είναι αυτή της αλλαγής του κλίματος. Στη βάση αυτού του σενάριου που ε, μας έφερε μέσα σε λίγα χρόνια από την αυθονία στη Σπάνιδα είναι πολύ σημαντικές, αλλά υπάρχει και μια πολύ σημαντική ανισορροπία που δημιουργείται μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τα μοντέλα κατανάλωσης των πολυπληθών περιοχών του κόσμου που τις αποκαλούμε αναδυόμενες αλλάζουν και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση με εκθετικό βαθμό, σίγουρα πολύ μεγαλύτερη της ε, προσφοράς. Ο καθηγητής Πρόντι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το προφίλ του στο διεθνές προσκήνιο και πολλές φορές βρέθηκε στην ηγεσία πολύ σημαντικών πρωτοβολιών, κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο συμμετείχε και στο China Europe International Business School. Σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες θα, όπως θα μας επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο κύριος Πρόντι, υπήρχε πολύ ε, σημαντικό ενδιαφέρον για την ε, επισητιστική ασφάλεια, κυρίως για τη διάθεση και την εποχικότητα των προμηθειών και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη τροφίμων στις φτωχότερε χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή διευρύνεται και υπάρχουν πολύ σημαντικές ε, νέες συνιστώσεις που σημαίνει ότι πρέπει από κοινού να βρούμε μία λύση σε διεθνές επόπεδο. Σήμερα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συζήτηση και στο G20 και ίσως στο μέλλον μπορεί να έχουμε μια global full policy, αυτό το οποίο εύχομαι προσωπικό σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα καθηγητά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας εξ ονόματο όλων των ομάδων της, επιτροπή της Επιτροπής ε, Γεωργίας σε μια πολύ σημαντική στιγμή που αφορά ιδίω το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλου για την παρουσία σα και σα δίνω το λόγο κύριε Πρόντι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, μετά από πέντε χρόνια έρχομαι εδώ με ιδιαίτερη συγκίνηση. Δέχτηκα πολύ ευχάριστα την ε, πρόταση του κυρίου Ντεκάστρο να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις για το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα μαζί με το πρόβλημα της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης είναι αυτό. Πρόκειται για τρεις προοπτικές οι οποίες είναι αλληλένδετες και μας δίνουν και μια αίσθηση της ανάγκης να έχουμε νέες πολιτικές ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Η επιστημιστική ασφάλεια είναι αυτή που συζητάτε λιγότερο από τα τρία θέματα, αλλά κατ' και το πιο σημαντικό από όλα, διότι βρισκόμαστε σε μία καμπή. Βρισκόμαστε σε μία καμπή σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω το γεγονός ότι σήμερα είμαστε περίπου 7 δισεκατομμύρια αυτούς τους μήνες ε, θα φτάναμε λογικά στα 7 δισεκατομμύρια στον πλανήτη μας. Στα μέσα του αιώνα θα βρισκόμαστε στα 9 δισεκατομμύρια. και έχουμε μια ανάπτυξη λίγο κατώτερη από αυτή που περιμέναμε πριν από κάποια χρόνια μεν, αλλά υψηλότερη από αυτές που είχαμε στις ε, τελευταίες ε, προβλέψεις. Για να ε, σας εξηγήσω λίγο σαφώστερα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η αύξηση είναι 220.000 νέοι άνθρωποι κάθε μέρα. Αυτό σας δίνει μια εικόνα της τεράστιας πρόκλησης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από αυτούς ε, τα 2 δισεκατομμύρια και αν δεν παρέμβουμε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζουν με κάτω των 2 δολαρίων την ημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική αυτή είναι η ανάγκη. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία ε, αυξανόμενης αστικοποίησης. Το ίμιση περίπου του πληθυσμού του πλανήτη ζει στις πόλεις και το 70% θα ζει στις πόλεις ε, στα μέσα του αιώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το επισητιστικό πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής, είναι και θέμα επιμελητίας και θέμα στατιστικών και θέματα διατήρησης των αποθεμάτων. Όλα αυτά σημαίνουν και μεγαλύτερη ζήτηση σε τρόφιμα για διατροφικούς λόγους, πολύ περισσότερες ζωοτροφές για τα ζώα και ανάγκη όλο ένα και αυξανόμενης γεωργικής παραγωγής. Και επίσης σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση το εμπόριο των διατροφικών προϊόντων γίνεται πιο ελεύθερο και η ηρωνία της τύχης όμως ε, το κάνει και πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε, διότι δημιουργήθηκαν νέες προκλήσεις και δημιουργούνται συνεχώς νέες προκλήσεις και υπάρχουν και ανησυχίες για την επισητιστική ασφάλεια. Εδώ και κάποια χρόνια για κάποιες χώρες, για να ξεκινήσουμε από την Κίνα που είναι η πιο προφανής, αλλά επίσης και για την Ινδία, το πρόβλημα της επισητιστικής ασφάλειας είναι πλέον ένα ρητό στρατηγικό πρόβλημα της εθνικής πολιτικής. Μια απόλυτη προτεραιότητα της εθνικής τους πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι μια περαιτέρω πρόκληση είναι η διακύμανση των αγορών, δηλαδή επειδή υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στις οικονομικές ροές και στην κατάσταση των αγορών, στα ποσοστά αλλαγής ε, ε, συναλλάγματος και στην αλλαγή της τάσης των καταναλωτών για την ποιότητα. Επίσης υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με τις τεχνολογικές πρόοδους του τομέα. Εμείς ακόμα δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις όσον αφορά τα θέματα της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας, ε, της ε, ε, λεγόμενης επακριβούς γεωργίας, της γεωργίας της ακρίβειας. Πρόκειται για τομείς που είναι αλληλένδετοι με τα προβλήματά μας. Και τέλος, υπάρχει και η εξής πρόκληση. Ποιος πληρώνει το τίμημα για τα δημόσια αγαθά που παράγονται αγαθά τα οποία δεν πληρώνει η αγορά. Όπως για παράδειγμα η ύπεθρος, ε, η συντήρηση του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική προστασία, η βιοποκυλότητα. Όλα αυτά είναι αντικειμενικές υπηρεσίες προς την ανθρωπότητα, οι οποίες ε, είναι αλληλένδετες με τον πολιτισμό μας, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να πληρώσει με τις τιμές της αγοράς enorme, è un problema di Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα λοιπόν. Και υπάρχει σπάνιδα και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο. Διότι αυτή τη στιγμή εξαντλούνται σχεδόν σε όλο τον κόσμο οι δάτινοι πόροι, οι υδροφόροι ορίζοντες, το νερό χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για αστική κατανάλωση και αυτό φυσικά μας οδηγεί σε απώλειες ε, στο έδαφος και στην ε, ε, δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το νερό για παραγωγή διατροφικών προϊόντων. Φυσικά γίνεται η σύνδεση του ύδατος με τα τρόφιμα, διότι η έλλειψη νερού μεταφράζεται και σε έλλειψη τροφίμων. Ενώ εμείς κάθε μέρα καταναλώνουμε από 2 έως 4 λίτρα νερό, χρειαζόμαστε 2 λίτρα νερό ημερησίως για την παραγωγή των τροφίμων που καταναλώνουμε και χρειαζόμαστε περίπου ένα λίτρο νερό για κάθε θερμίδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και των ε, υδάτινων χρήσεων παγκοσμίω είναι για τη γεωργία. Και η επανάσταση αυτή δεν είναι μόνο δημογραφική, πρόκειται και για μια επανάσταση στον ε, τύπο της διατροφής και το πέρασμα από τις πρωτεΐνες σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες, ε, περισσότερα εδάφη. Ξέρετε ότι για να έχουμε ένα χιλιόγραμμο κρέατος χρειαζόμαστε περίπου 8 χιλιόγραμμα δημητριακών που σημαίνει ότι ε, χρειαζόμαστε 8.000 λίτρα νερού για την παραγωγή τους. Υπάρχουν και άλλοι ε, παράγοντες βέβαια, όπως ε, η υπερεκμετάλλευση των εδαφών, ιδίω σε περιοχές όπου δεν επιτρέπει η φυσική ε, δομή του εδάφους να το χρησιμοποιούμε και θα πρέπει να γίνουν και κάποιες μετατροπές ή επίσης η χρήση των βιοκαυσίμων, που είναι ένα από τα ουσιαστικά προβλήματα. όταν δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός ε, και υπήρχε η απόλυτη ευθυμία του εδάφου σε σχέση με τη ζήτηση, δεν υπήρχε και πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τίθεται το πρόβλημα και μάλιστα είναι και από τα πρωταρχικά. Οι καλλιεργητές προσπαθούν να εξισορροπήσουν τη ζήτηση και την προσφορά τροφίμων Τίθεται το πρόβλημα πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον και όλα αυτά είναι ε, στοιχεία που εξετάζουμε από κοινού. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος απευθείας και θα πρέπει καταρχάς να θέσουμε και το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ ενέργειας και τροφίμων για τη χρήση των εδαφών. Δεν έχω καμία αμφιβολία λοιπόν ότι στον ανταγωνισμό μεταξύ τροφίμων και ενέργειας θα πρέπει να επιλέξουμε κατά προτεραιότητα τα τρόφιμα. Βεβαίως, είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες εκμετάλλευσης των γεών παγκοσμίω. Υπάρχουν καινοί χώροι στη γη που προσελκύουν την προσοχή όλων ε, παγκοσμίω, ε, ιδίω αυτών που έχουν ε, ανάγκη τροφίμων, όπως είναι η Αφρική και η Λατινική Αμερική και εκεί επικεντρώνεται και μεγάλο τμήμα του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι νέε γέ βέβαια δεν είναι επαρκής και σε πολλές περιπτώσεις είναι και ακατάλληλες διότι πρόκειται για εδάφη δεύτερης κατηγορίας που είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν για διατροφική χρήση και σε πολλές περιπτώσεις περιπλέκονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα διότι υπάρχουν αμφίσιμες καταστάσεις ως προς την ιδιοκτησία και τη χρήση των γεών. Και επίσης επειδή δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες κυβερνητικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές, αυτά τα νέα εδάφη, αλλά η μεγαλύτερη προσπάθεια θα πρέπει να είναι, να είναι πιο παραγωγικά αυτά τα εδάφη τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν, τα νέα συστήματα άρρωσης, οι νέες τεχνικές καλλιόργειες που απαιτούν λιγότερη ενέργεια, αλλά οι νέες τεχνολογίες αποδεικνύουν τη συνδρομή τους μέχρι ενός σημείου. Διότι υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου, δεδομένου ότι πρόκειται και για μια εκβάθρον αλλαγή, και αυτό είναι το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες που αυξάνουν την ε, παραγωγικότητα του εδάφους ε, τα τελευταία χρόνια ε, φθήνουν και έχουμε φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και στα όρια της αποτελεσματικότητας της φωτοσύνθεσης. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά προβλήματα αν θέλουμε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα. Για να ε, σας δώσω μια εικόνα του πόσες είναι οι αλλαγές στον κόσμο, Στι προσπάθειες που γίνονται και στις αλλαγές ε, των προϊόντων ανά στην Ινδία, στην ε, Κίνα, στη Ρωσία ε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να, αναστρέψουμε τη μείωση στην παραγωγικότητα της γεωργίας η οποία ήταν κατά 4% στη δεκαετία του 60-70 μέχρι και τη δεκαετία του 80 και αυτή τη στιγμή σύμφωνα και με τις προβλέψεις για το 2030 ε, μόλις και με τα βίας φτάνουμε στο 1%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ έχουμε αλλάξει. Έχει αλλάξει η παραγωγικότητα από το 4% στο 1% που σημαίνει ότι έχουν αλλάξει εκβάθρων οι προοπτικές μας. Και αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και εισαγωγέας τροφίμων και ο ρόλος μας ως προμηθευτής τροφίμων παγκοσμίων φθήνει συνεχώς. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης των 27 στο μέλλον σίγουρα θα επιδεινωθεί ή τουλάχιστον όλες οι προβλέψεις λένε ότι υπάρχει πιθανή επιδείνωση για κάποια δημικριακά, μάλιστα για το σιτάρι η Ευρώπη από καθαρός ε, εξαγωγέας θα γίνει καθαρός εισαγωγέας. Και ακριβώς ε, η χρήση των εδαφών που κάναμε για ενεργειακούς σκοπούς είναι τμήμα της ευθύνης μας. Η δυνατότητα της Ευρώπης λοιπόν να αντιμετωπίσει την ένδια παγκοσμίω είναι κάτι το οποίο μειώνεται συνεχώς. Η κατάσταση αυτή βέβαια στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο διαφορετική από την κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείε, διότι και στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα χρήσης των γεών, ιδίω των καλύτερων εδαφών για ενεργειακούς σκοπούς και επομένως πρόκειται για κοινό πρόβλημα για τις χώρες που έχουν υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Το θέμα των τιμών πριν από τρία χρόνια ήταν σαφέστατο παράδειγμα. Μετά μειώθηκε όλο ε, το θέμα της αύξησης των τιμών. Δεν είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής όπως ήμασταν πριν από τρία χρόνια, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους παρισταμένους ότι η επιστημιστική κρίση θα ξανάρθει, διότι τα στοιχεία της ανάπτυξης και οι επιστημονικές προβολές καταδεικνύουν ότι ε, φτάνουμε προς την έλλειψη να μην ξεχνάμε δε ότι αν δεν αλλάξουμε πολιτικές και αν συνεχίσουμε με τη σημερινή πολιτική θα φτάσουμε σίγουρα στην έλλειψη. και δικαίω μας εκρούει τον κόδυνα του κινδύνου η ΦΑΟ, διότι θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την αίσθηση ασφάλειας και να μην λησμονούμε ότι πριν από τρία χρόνια φτάσαμε σε τεράστια γεωργικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα, όπω ανέφερα προηγουμένως, σαφείς ενδείξεις ότι γίνεται μια παγκόσμια μάχη πλέον για τα τρόφιμα και ιδίω για πρώτη φορά στην ιστορία ε, γίνεται μία μάχη για τις αρρώσιμες εκτάσεις που παράγουν ε, τρόφιμα. Το συζητήσαμε και όπως ε, αναφέρει και η ΦΑΟ έχουμε πλέον νεοαπικιακές τάσεις. Ε, όλο ένα και αυξανόμενο αριθμό χωρών, η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία, όλε οι χώρε του κόλπου αρχίζουν να αγοράζουν εκτάσει με μακροπρόθεσμε συμβάσει ή με διάφορε μορφέ αγορά εκτάσεις στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού ε, αντιμετωπίζεται δυσκολία. Δεν είναι ίσονο σημασία στο πρόβλημα. Λέγεται ότι υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις για πάνω από 60 εκατομμύρια εκτάρια. Αυτό είναι μεγαλύτερο της ε, ε, αρρώσιμης επιφάνειας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας μαζί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πλέον στρατηγική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική στρατηγική τεραστίων διαστάσεων. Αυτή η μάχη για τις αρρώσιμες γέες κατεδεικνύει πόσο σημαντικό έχει γίνει το πρόβλημα της ε, επισητιστικής ε, ασφάλειας. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ε, παρισταμένους για να τους ευαισθητοποιήσω και λίγο από πολιτική σκοπιάς, να φανταστούν τι μπορεί να προκύψει και τι προβλήματα μπορεί να ανακύψουν εάν μία αφρικανική χώρα στην οποία εκατομμύρια εκτάρια δίνονται προς εκμετάλλευση σε αλλοδαπούς βρεθεί ξαφνικά σε κατάσταση έλλειψης τροφίμων. Φανταστείτε αυτό την εκδοχή που δεν είναι μια αφηρημένη εκδοχή, είναι κάτι το οποίο είναι καθόλου πιθανό και να σκεφτούμε λίγο ποιες είναι οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Δεν θα, θα αναφερθώ βέβαια εδώ σε παράπλευρες πτυχές. Ε, στην αρχή σας ανέφερα ότι είναι αλληλένδετη η περιβαλλοντική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση και η επισητιστική κρίση ε, και για την κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη σχέση της με την επισητιστική ασφάλεια είναι σαφές ότι το γεγονός ότι τα κονδύλια που μειώνονται για τη γεωργία, οι δυσκολίε της πιστώση έχουν δημιουργήσει αντικειμενικές δυσκολίε και στη γεωργία. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό το σημείο, αλλά να το έχετε κατά νου, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν σήμερα, για να ολοκληρώσω με αυτή τη στοιχή, σε αυτό το πρώτο τμήμα της παρέμβασής μας, υπάρχει ισορροπία, και μια κάποια ισορροπία στις αγορές ακόμα, είναι γιατί υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας και άλλο ένα δισεκατομμύριο που βρίσκονται κάτω από το κατάφλι των δύο δολαρίων την ημέρα. Καταλαβαίνετε πόσο πιο έντονα είναι τα προβλήματα από αυτό που φανταζόμαστε. Βεβαίως, πέραν της πτυχής της ασφάλειας, προκύπτει απευθείας και το θέμα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. διότι αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή μετά από την στοιχειώδη πτυχή της ασφάλειας. Για πολύ μεγάλο διάστημα η περιβαλλοντική ασφάλεια είναι η εικόνα, η προβολή της επισητιστικής ασφάλειας. Διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τρόφιμα αν δεν έχουμε καθαρό νερό, αν δεν υπάρχουν αρρώσιμες γιές, αν δεν υπάρχουν κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και συνεπώς η έλλειψη μιας περιβαλλοντικής πολιτικής και η επιδείνωση του περιβάλλοντος διακυβεύουν φυσικά και την γεωργική παραγωγή. Και φυσικά θα πρέπει να παρέμβουμε και σε αυτό το τομέα. Πρέπει να κάνουμε μία απόπειρα, να έχουμε μία γεωργία που θα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, επιστημονικές δομές ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό και Παραδείγματο χάρη με τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και πάρα πολλέ άλλε διαδικασίε, τεχνολογία. Ε, δίνεται εντύπωση ότι η τεχνολογία θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τουλάχιστον τις ζημίες από τα ε, πολύ αλμυρά ύδατα, πολύ αλμυρές εκτάσεις και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εκτάσεις που αυτή τη στιγμή δεν είναι καλλιεργήσιμες. Και φυσικά να δώσουμε και κάποιες λύσεις και να μην δημιουργήσουμε χειρότερες καταστάσεις. Θα πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου το εξή. Η έρευνα και η ανάπτυξη στο γεωργικό τομέα παγκοσμίως μειώνονται συνεχώς στην τελευταία γενιά. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή αυτή η γενιά που έχει αυτή την ψευδέστηση της ασφάλειας εμπιστεύτηκε και θεώρησε ότι, τη Γεωργία και θεώρησε ότι πρέπει η παγκόσμια έρευνα να γίνει προς άλλες κατευθύνσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πρόοδοι ε, και σας ανέφερα και κάποιες, αλλά είναι πολύ αργές, διότι δεν υπάρχει αίσθηση της προτεραιότητας και της κρίσιμης κατάστασης της γεωργίας. Και θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω αυτό, διότι κατ' εμέ είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγαλύτερο σθένος στην ε, μελλοντική μας πολιτική. Σας υπενθύμισα λοιπόν τα στοιχεία αυτά, διότι Εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την πολιτική μας και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας συνεχώς προκειμένου να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές είτε τις ε, αυστηρά παραγωγικές είτε τις παραγωγικές και παραβολητικές πτυχές της γεωργίας. Ζαφώς ανακύπτει και ένα ακόμα πρόβλημα και εδώ φτάνω και προς το τέλος της παρέμβασής μου Εάν εμείς θέλουμε η γεωργία να είναι ενεργή στην παραγωγή των δημοσίων αγαθών, δηλαδή να ε, είναι φιλική προς το περιβάλλον, να μην υπάρχει επιδείνωση ε, του περιβάλλοντος χώρου, όλα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να λάβουμε υπόψη και αυτό αυτή την πτυχή της γεωργίας. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, διότι το παρόν σύστημα τιμολόγησης δεν λαμβάνει υπόψη το αυτή την πτυχή. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει και αύξηση της ηλική παραγωγής για κάποιο διάστημα, αλλά αν δεν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο για την ε, αποσμίωση και των δημοσίων αγαθών που μας δίνει η παραγωγή τροφίμων, αναπόφευκτα θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Και εδώ φυσικά επαφείται στην ε, πολιτική, στην πολιτική των επιδοτήσεων και της βοήθειας. Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική επιδετήσεων που δεν θα προκαλεί στρεβλώσεις. Οποιαδήποτε επιδότηση προς τη γεωργία, οποιαδήποτε προσοχή προς τη γεωργία δεν ε, μπορεί παρά να οδηγήσει στη μείωση της προσοχής μας ε, για τα δημόσια αγαθά. Πρόκειται λοιπόν για ένα οικονομικό άχθος ιδιαίτερα άμεσο. Μία από τις τελευταίες πτυχές που θα ήθελα να θίξω τώρα είναι το θέμα της διαχείρισης των παγκοσμίων αγορών γεωργίας. Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε μία ε, πόλωση στα συναισθήματα και στη διανόηση. Κάποιοι θεώρησαν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ο τελευταίος παράδεισος επιγής, ότι το εμπόριο μας οδηγεί στην ευτυχία και τα πράγματα είναι τέλεια. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για απάτη που στερεί θέσεις εργασίας και ότι γίνεται μόνο προς όφελος των κερδοσκόπων. Και έτσι ο κόσμος βρίσκεται διαιρεμένος και αυτή η διχογνωμία καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει μία παγκόσμια διακυβέρνηση σε γεωργικό επίπεδο. Και θα πρέπει να το αναλογιστούμε το συγκεκριμένο γεγονός, διότι αυτό είναι και αυτό που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, στον ε, ΠΟΕ, στον κύριο της Δόχα. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες ρίζουν, ε, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ στεναρές οι απόψεις εκατέρωθεν, δεν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης και σε διεθνές επίπεδο πλέον παραμένει το πρόβλημα, διαιωνίζεται εδώ και χρόνια και δυστυχώς προσωπικά φρονώ ότι δεν μας μένει και πολύ καιρό ε, για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Ε, προσωπικώς υποστηρίζω την παγκοσμιοποίηση, θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη για παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν πιστεύω και σε μία ε, φρενήρη πολιτική η οποία δεν έχει κανένα σταματημό. Διότι η αγορά αναμφίβολα μας βοηθά να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας, αλλά εάν δεν γίνεται με τα κριτήρια που σας υπενθύμισα προηγουμένως, σίγουρα θα φτάσουμε ένα σημείο όπου και η ίδια αγορά θα σταματήσει και δεν θα μπορεί να προχωρήσει άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολύ πιο υπεύθυνη θέση παγκοσμίω ε, για το εμπόριο, προκειμένου να αποφύγουμε να μας οδηγήσει η μαγκοσμιοποίηση στο να έχουμε πιο πλούσιους ανθρώπους, να μειώσουμε την ένδυα των ε, ε, περισσότερων και παγκοσμίω να οδηγηθούμε στη στασιμότητα. Όπως σας έλεγα, ο γύρος της Δόχας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν γίνει μία πλήρης αλλαγή της παγκόσμιας κυβέρνησης, της governance. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, ε, θα μπορούσαμε ίσως να αναφέρουμε κάποια στοιχεία στη διάρκεια της συζήτησης αργότερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια εντονότατη ασυμμετρία αυτή τη στιγμή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις, παγκο... τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Οι αναπτυγμένες χώρες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ πιο εύκολα την ε, απελευθέρωση, διότι μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα, διότι έχουν περισσότερους πόρους για να μπορέσουν να κινηθούν, ενώ οι χώρες ε, οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες βρίσκονται σε πολύ πιο μειονεκτική θέση αυτή τη στιγμή και δυστυχώς χρειάζονται και χρόνο και πόρους, πολύ περισσότερο από εμά ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή εισοδεύουμε προς την παγκόσμια σπάνιδα των τροφίμων. Είναι αναμονόμενη και η έλλειψη συμμετρίας μεταξύ των χωρών που έχουν υπερβολική παραγωγή και των χωρών που είναι εισαγωγής. Να σας πω το εξής τα τελευταία χρόνια της ιστορίας μας δεν είχε διαπιστωθεί ποτέ να υπάρχει απαγόρευση ή περιορισμός στην εξαγωγή διατροφικών προϊόντων. Ήταν περιορισμένη διάρκεια βέβαια, περιορίστηκε σε κάποιες και μένων χώρων, αλλά πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό σήμα κινδύνου διότι τούτο σημαίνει ότι αφενός υπάρχει παγκοσμιοποίηση, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να διακόψουμε την παγκοσμιοποίηση ε, άξαφνα μόλις έρθει η έλλειψη. Το γεγονός ότι η Ρωσία, η Αργεντινή και άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια είτε περιόρισαν είτε απαγόρευσαν κάποιες εξαγωγές είναι ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την απεσιόδοξη ανάλυση που σας έκανα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες επανήλθαμε σε ε, δελτία, ενώ οι χώρες οι οποίες έχουν κάνει ε, περιορισμούς έχουν την εντύπωση ότι έτσι θα μειώσουν την παγκόσμια έλλειψη τροφίμων, ενώ στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα ε, κυκλικό φαινόμενο που θα επηρεάσει τους πάντες. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατάσταση, να λειτουργήσουμε με σοφροσύνη στις επιδοτήσεις μας διότι όπως σας έλεγα και πριν αν κάποιος απαγορεύσει απευθείας τις επιδοτήσεις διότι θεωρεί ότι έτσι θα έχουμε εξυγίανση του γεωργικού τομέα οι χώρες οι οποίες ε, είναι καθαρή εισαγωγή τροφίμων θα πληχθούν περισσότερο διότι με την κατάσταση που σας περιέγραψα θα έχουμε μία απότομη αύξηση των τιμών και θα υπάρχουν προβλήματα. Ενώπιον αυτής της κατάστασης βρισκόμαστε, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, διχογνωμίες μεταξύ των χωρών και υπάρχουν και διακυμάνσεις των τιμών οι οποίες θα αυξάνονται συνεχώς. Αυτές είναι λοιπόν οι προοπτικές που έχουμε ενώπιόν μας. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι η αγορά έχει ενδιαφυσβήτητα Άσε αυτή την άποψη ότι με το μαγικό ραβδάκι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις και αυτή είναι η απέτηση όλων. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν στρεβλώσεις, αυτό είναι σαφές, αλλά η ιδέα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ίχνος γεωργικής πολιτικής παγκοσμίω είναι σίγουρα εσφαλμένη χρειαζόμαστε γεωργικές πολιτικές οι οποίες θα είναι αρρωγός του παγκοσμίου εμπορίου αλλά κυρίως θα είναι και πολιτικές οι οποίες θα φροντίζουν το πρόβλημα του περιβάλλοντος και της έλλειψης στις φτωχότερες χώρες. Ολοκληρώνοντας, να σας πω το εξής. Χρειαζόμαστε καταρχά μέχρι το 2050 να διπλασιάσουμε την παγκόσμια γεωργική παραγωγή, διότι θα γίνουμε από 7, 7 δισεκατομμύρια 9 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να υπάρχουμε ε, διατροφικές δυνατότητες για να καλύψουν περισσότερα προϊόντα, άρα και μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Παρένθεση εδώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη και στην ε, τεράστια κατασπατάληση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Η λόγω συγκεκριμένων συνηθιών των ε, ε, καταναλωτών ή και για την ε, ενέργεια για το κρύο ή για την έλλειψη κρύου γίνονται τεράστιες σπατάλες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη να σκεφτούμε το μέλλον μας και να εκπονήσουμε μία πολιτική την οποία θα σας την παρουσιάσω επιγραμματικά με δύο-τρία σημεία. Καταρχάς πρέπει να αυξηθεί η τάση της παραγωγικότητας στη γεωργία. Δεν το επισημαίνει κανείς ποτέ, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο σημείο. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο επίπεδο για να ξεκινήσει επίσης εκ νέου η έρευνα και η ανάπτυξη στη γεωργία. Να δημιουργήσουμε τις τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις ώστε να διαδοθούν οι καινοτομίες σε όλο τον κόσμο. Και μόνο διότι η γαλλική, η γερμανική, γεωργία μπορεί να γίνουν πιο αποτελεσματικές, αλλά γιατί θα πρέπει να διαδοθούν ταχύτατα οι καινοτομίες. Δεύτερον, τα τρόφιμα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Η διατροφή είναι προτεραιότητα. Θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα λοιπόν ώστε να δοθούν κίνητρα για τη γεωργική παραγωγή, να μην τα δώσουμε στη μη γεωργική προεγωγή και να φροντίσουμε και να μην δίνουμε αρρώσιμες εκτάσεις για άλλους λόγους. Η, τα τρόφιμα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε επί πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. Αυτό που σας είπα πριν για τις ερώσιμες εκτάσεις είναι πολύ σημαντικό και δεδομένης και της διαδικασίας της μελλοντική αστικοποίησης θα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων αποτελεσματικά η χρήση της γης ε, στη νέα αστική πολιτική. Το πρόβλημα της ανάκτησης, το πρόβλημα της εξοικονόμησης εδαφών θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ενώ η τελευταία γενεά ήταν ε, ε αυτή που έθετε το ζήτημα ως δευτερεύον. Τρίτον, ή μάλλον τέταρτον, χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση του ύδατος ήγηκε πλέον η στιγμή να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία. Τα συστήματα ίδρυυσης τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι ε, συστήματα τα οποία είχαμε δημιουργήσει όταν ήταν ελεύθερο αγαθό το νερό και δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ανανεώσουμε πλήρως τις τεχνολογίες μας και αυτό δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι πρόβλημα ειρήνης ή πολέμου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους παρισταμένους τι γίνεται στου μεγάλου ποταμού του κόσμου. Να σα δώσω το παράδειγμα του, Νίλη, το, του το ίδιο ισχύει και για τον Τίγρη και τον Εφράτη και του Αμερικανικού ποταμού και τον... και τα αφρικανικά ποτάμια. Τα νερά είναι σχεδόν τα ίδια. Φτάνουν στη Μεσόγειο σχεδόν ε, ξερά πλέον τα ποτάμια, ξηρά, είναι ελάχιστη η υδροδότηση και υπάρχουν ε, ε, στον ήλο μεταξύ, με παλιές συνθήκες που υπάρχουν μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου. Πλέον η Αφρικανικέ χώρε ζητούν μεγαλύτερη χρήση του νερού. Το Σουδάν έγινε πλέον δύο χώρε. άρα υπάρχουν διαφορετικέ κατανομές. Σα εφιστώ την προσοχή, πρόκειται για καταστάσει οι οποίε θα γίνουν πάρα πολύ κρίσει. Ό,τι συμβαίνει στον Ήλο θα γίνει και σε άλλα ποτάμια. Και αυτή τη στιγμή με χρήση των τεχνολογιών που έχουμε αυτή τη στιγμή, με πιο σύγχρονες τεχνολογίες θα είχαμε καλύτερη χρήση του ύδατος και με καλύτερη χρήση ε, θα έχουμε ε, καλύτερες λύσεις και είναι μικρές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν αλλά χρειαζόμαστε διεθνή προγράμματα διότι θα τεθεί το ζήτημα της ειρήνης του πολέμου και της έλλειψης νερού για όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία ήθελα να σας θέσω. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι στα μέτρα μας, διότι έχουμε και άλλες πηγές ενέργειας πλέον. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές, δεν εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές, θα βρεθούμε ενώπιον μιας γενικότερης και απαράδεκτης αύξησης των τιμών και σας επαναλαμβάνω αυτό θα γίνει σε πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα διότι η ζήτηση των τροφίμων αλλάζει ταχύτατα και αλλάζει και η παγκόσμια ισορροπία. Δεν αναφέρομαι σε 20 χρόνια μετά, αναφέρομαι σε λίγα χρόνια μετά. Επομένως πρέπει να κινητοποιηθούμε, να γίνει μια παγκόσμια ενωμένη προσπάθεια για να αντιμετωπιστούμε στις μεγάλες προκλήσεις και να προσφέρουμε τρόφιμα σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε πάρα πάρα πολλά ερεθίσματα τα οποία ουσιαστικά αυξάνουν την ευθύνη της Επιτροπής μας, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου. Και αυτές τις μέρες βέβαια με την έκθεση ΔΕΣ ουσιαστικά θα δώσουμε και εμείς ένα όραμα για το μέλλον της πολιτικής αυτής. Και δεν μπορούμε παρά να μην λάβουμε, παρά να λάβουμε υπόψη μας την δραματική αυτή η κατάσταση την οποία περιγράψατε, η οποία θα μας απασχολήσει πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε. Πρέπει λοιπόν πολύ γρήγορα και εκ του σύνεγγυς να ασχοληθούμε με την κατάσταση αυτή. Κύριε καθηγητά, ο συνήθως θα δώσουμε τώρα τον λόγο πρώτα στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσετε και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο του χρόνου προκειμένου να ακούσουμε και ερωτήσεις από τους άλλους βουλευτές που είναι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και ξεκινάμε αμέσως με τον συντονιστή του ΕΛΚ, που είναι και εισηγητής της έκθεσής μας, ο κύριος Ντες Άλμπερτ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητά, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ακούγοντας ε, την ομιλία σας, ε, κύριε καθηγητά, διαπιστώνω ότι διαβάσατε τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Πολλά από αυτά που θα αποφασίσουμε, ελπίζω τουλάχιστον σήμερα το απόγευμα, μετά από συζήτηση των τροπολογιών μας, τα θίξατε τα συμπεριλάβατε σε αυτά που είπατε, όπως παραδείγματο χάρη τη συμβιβαστική τροπολογία 2 που αναφέρεται στην επιστηστική ασφάλεια, που είναι ουσιαστική για εκατομμύρια άτομα και στην Ευρώπη. Θεωρούμε πραγματικά ότι και η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό. Μιλήσατε επίσης ε, και στις επιφάνειες. Μιλήσατε επίσης και για τις επιφάνειες ε, λέγοντας ότι πραγματικά η δημογραφική ανάπτυξη είναι κάτι που μας απασχολεί. Ελπίζω πραγματικά ότι οι μεγάλες ε, επιφάνειες γης οι οποίες έχουν αποσυρθεί από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων θα επανέλθουν και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε καθηγητά γιατί πραγματικά με θάρρος αναφέρετε τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο και εμείς για την θέση των ε, αγροτών στην Ευρώπη, για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων βασικών και απαραίτητων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η γεωργία στην Ευρώπη η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε με την γνωστή ρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής με τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα και με τις δυνατότητες που είχαν οι αγρότες να μην παράγουν και να λαμβάνουν κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι Οι πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά την αγορά, την εξαγορά επιφανειών γης ε, από Κινέζους στην ε, ε, πληροφορία αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγνοήσουμε και έχω την εντύπωση ότι η εξαγορά επιφανειών γης στην Αφρική παραδείγματο χάρη από Κινέζου. δεν πρόκειται για χρησιμοποίηση, για εκμετάλλευση, πρόκειται για αγορά. Είναι κάτι που σαφώς και θα πρέπει να μας αποσχολήσει. Το θέμα της στόχης στον τρίτο κόσμο διαθέτουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επιδοτήσεις στις εξαγωγές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν αφορο τις οποίες δεν αφορά το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν περισσότερο στην πολιτική μας. Εγώ έχω πάει σε πολλές χώρες της ε, Αφρικής, ε, μάλιστα έχω και μέλη της οικογένειάς μου που ζουν εκεί. Και παραδείγματος χάρη η Ροδεσία, σήμερα Ζιμπάμπουε, ήταν ε, ένας από τους σημαντικούς προμηθευτές σιταριού του κόσμου και σήμερα η κατάσταση είναι δραματική πεινάνε οι άνθρωποι που ζουν σήμερα στην περιοχή αυτή και είμαστε εν μέρη υπεύθυνοι. Μιλήσατε βεβαίως και για τις σχέσεις μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος και έχετε δίκιο ότι είναι σήμερα πολύ σημαντικό να ξαναδούμε το φαινόμενο αυτό. Βεβαίως και υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο αυτών τομέων και όταν μιλάμε για την αηφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται η έννοια της ε, αηφόρου ανάπτυξης είναι κάτι που βεβαίως σε μεγάλο βαθμό αφορά και τις ε, δασικές ε, επιφάνειες, τις δασικές εκτάσεις. Οι περισσότεροι αγρότες στο παρελθόν προσπαθούσαν να μεταβιβάσουν τις περιουσίες τους στα παιδιά τους. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου που αυτό δεν μπορεί να γίνει, όπου δεν είναι βιώσιμη αυτή η δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω και εγώ ότι τα περισσότερα από τα θέματα που θίξατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και γι' αυτό και θα ήθελα να μιλήσω και για την τροπολογία 49 όπου μιλάμε βεβαίως για την ρύθμιση των αγορών, τους μηχανισμούς δηλαδή που θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους αγρότες να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς ρύθμισης και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γεωργούς στην Ευρώπη οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν κάποια αποζημίωση. Δεν πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι κάτι το απαραίτητο για να στηρίξουμε την παραγωγή στην Ευρώπη. Θα ήμουν ευγνώμων αν μας πείτε όταν ξαναπάρετε το λόγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Σαρκοζής, το G20, έχουν έχει συμπεριλάβει το θέμα των πρώτων υλών, των βασικών γεωργικών προϊόντων, καθώς και της κερδοσκοπίας, αναφέρει τις τιμές των πρώτων υλών. Και βεβαίως ε, ότι θα πρέπει να ανοίξει η ευρωπαϊκή αγορά στα προϊόντα αυτά τα οποία προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρετε ποια είναι η πολιτική της Αμερικής και άλλων περιοχών για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρώτη για τα περισσότερα από όσα είπατε. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πλήρως σύμφωνος. Ευχαριστώ πολύ. Άλμπερτ. Ευχαριστώ και όλους όσους είναι εδώ, παρόντες. Και θα δώσω μέσω το λόγο στον Λουίς Καμπούλα Σάντος, ο οποίος είναι επίσης ε, συντονιστής για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα ήθελα να πω ότι είναι καταρχάς πολύ μεγάλη τιμή που σας έχουμε μαζί μας σήμερα κύριε Πρόντι σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε και εσείς στην ε, κρισιμότατη αυτή συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα θα λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εσείς, κύριε Πρόντι, Είστε μια προσωπικότητα πολύ σημαντική στον τομέα αυτό και μιλήσατε για τον ε, ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της επισητιστικής ασφάλειας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίω. Αναφερθήκατε σε στοιχεία, σε διάφορους τομείς οι οποίοι είναι τόσο πολιτικοί, τεχνικοί όσο και ιδεολογικοί. Είπατε επίσης ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο τα όσα μας μαθαίνει η τεχνολογία, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη γεωρική παραγωγή, πώς θα μπορούσαν να ρυθμιστούν οι ε, αγορές, οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Αντιμετωπίσουμε όμως ένα σημαντικό παράδοξο. Υπάρχει μια αντίφαση μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε ένα μοντέλο, ακολουθούμε αν θέλετε μία νοτροπία που βασίζεται στην συνεχή κατανάλωση και τη συνεχή παραγωγή. Βασιζόμαστε δηλαδή στην παραγωγή των προϊόντων αυτών που πολύ συχνά προέρχονται από κάποιες πρώτες ύλες οι οποίες δεν είναι ανανεώσιμες. Η παραγωγή αυτή, αν συνεχιστεί έτσι, θα είναι βράχη πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα μη βιώσιμη. Και ουσιαστικά εδώ πέρα χρησιμοποιούμε την μέθοδο εκείνη που παραδόξως τελικά χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή και οι αναδυόμενες οικονομίες, οι αναδυόμενες κοινωνίες. Αν αρχίσουν όλοι οι πληθυσμοί είτε, προ, είτε βρίσκονται στην Ινδία είτε βρίσκονται στην Κίνα, να χρησιμοποιούν όλοι μόνο αυτοκίνητα, θα βρεθούμε πολύ γρήγορα στην ίδια, θα βρεθούν και αυτοί στην ίδια δύσκολη κατάσταση που έχουμε κι εμεί. Αν αρχίσουν να καταναλώνουν τόσο πολύ χαρτί σαν αυτό το οποίο καταναλώνουμε στην Ευρώπη, θα ξεφανιστούν τα δάση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αναδυόμενες οικονομίες επιλέγουν το δικό μας δυτικό αναπτυξιακό μοντέλο και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο στο οποίο θα ήθελα να αφαιρθώ. Από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τις δικές μας μεθόδους κατανάλωσης, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα για τις υπόλοιπες οικονομίες, τις συναδειόμενες που τελικά υιοθετούν τις δικές μας μεθόδους. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για τη σφαιρική εικόνα την οποία μας δώσατε, για την κατάσταση όπως τη φωτογραφήσατε. φωτογραφίσατε. Οποιοδήποτε πολίτης που ανησυχεί για το μέλλον του πλανήτη θα συμφωνήσει προφανώς μαζί σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να μας πείτε κάτι παραπάνω για τη νέα τάξη πραγμάτων πόσο βιώσιμα θα είναι τα πράγματα στο μέλλον. Πιστεύετε κι εσείς ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης σαν αυτό το οποίο περιγράψατε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την παγκόσμια διακυβέρνηση την οποία εύχεστε. Ευχαριστώ. Nicholson, Το λόγο τώρα έχει ο Τζέιμς, συντονιστής ε, της ομάδας των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων, με συγχωρείτε. Σα e uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόντι για την παρουσίαση την οποία μας κάνατε εδώ πέρα. Εντοπίσατε κάποια πολύ σημαντικά σημεία, ενώ δεν είχατε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Όταν συναντάω γεωργούς αγρότες, Πολύ συχνά δημιουργείται το ερώτημα ότι δημιουργούμε τελικά πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και τελικά οι γεωργοί δεν έχουν μια απόλυτη ελευθερία για να παράγουν. Και όπως είπε και ο Άλμπερτ Ντες, όσον αφορά τις ε, διμερείς συμφωνίες, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή μια διμερή συμφωνία με το Μερκοσούρ. Οι δικοί μας οι αγρότες πρέπει να παράγουν βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και βάσει αυτών των προδιαγραφών παράγουν πολύ ποιοτικά προϊόντα. Και από την άλλη όμως εισάγονται και προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κατά την άποψή μου δεν είναι τα πιο ποιοτικά. Για παράδειγμα, βοδινό κρέα από την Βραζιλία, το οποίο δεν παράγεται βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που είναι πολύ πιο ψηλέ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό πλήγμα για τους δικούς μας τους αγρότες. Είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει βέβαια να προσφέρουμε τρόφιμα στον κόσμο, να ταΐσουμε τον κόσμο. Και ο Λουίς βέβαια αναφέρθηκε σε αυτό αναφερόμενο στον γύρο της Δόχα. Δεν άκουσα το πρώτο τμήμα της ε, παρουσίασής σας και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θέτω πάντω το ακόλουθο ερώτημα που ενδεχομένω να καλύψετε. Μήπω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο σύγχρονη τεχνολογία στην παραγωγή τροφίμων. Για παράδειγμα, αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου δεν είμαστε σε θέση να εισάγουμε από την Νότια Αμερική και τις Ηνωμένε Πολιτείες σόγια γενετικά τροποποιημένη ενώ η σόγια αυτή απαιτείται προκειμένου να τραφεί το ζωικό κεφάλαιο. Ξέρω, Ζωζέ Μποβέ, ότι εσύ δεν συμφωνείς με αυτό. Μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε με μια τέτοια στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ουσιαστικά εθελοτυφλούμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που χρησιμοποιεί τη μοντέρνα αυτή τεχνολογία και προχωρά μπροστά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Τζέιμς. Και τώρα εξ ονόματος των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων, η κυρία Πόλσον, η Αντιπρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόντι ιδιαίτερα. Σαφώς χρειαζόμαστε εδώ κάποια κίνητρα, ε, εξωτερικά θα έλεγα, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς προς τα που θέλουμε να πάμε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω σε ποια σημεία διαφωνώ με τον κύριο Πρόντι. Όσον αφορά τις ε, καλλιεργήσιμες επιφάνειες, παραδείγματο χάρη, έχω την εντύπωση ότι εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές επιφάνειες αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν με τις επιφάνειες που έχουμε διαθέσιμες και ας τις χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, ας κάνουμε μια καλύτερη χρήση αυτών των επιφανειών. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το πιο αποτελεσματικό. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Σάντος. Έκανα ένα ερώτημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια οικονομία η οποία απλώς παράγει και καταναλώνει, παραγωγή και κατανάλωση δεν μπορούμε να βρούμε και κάποιες άλλες μορφές ε, κατανάλωσης και κάποια άλλη μορφή παραγωγής. Μία βιώσιμη γεωργία η οποία θα μας εξασφαλίσει το μέλλον. Κύριε Πρόντι, μιλήσατε πολύ και για το νερό, μιλήσατε επίσης και για την υπερβολικά εντατική εκμετάλλευση της γης. Τι παράγουμε και πώς το παράγουμε. Βεβαίως όλα αυτά, εάν συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αποθέματα. Επίσης το θέμα της ενέργειας, από όπου προέρχεται η ενέργεια ως ε, ένα βαθμό. Δεν κοιτάμε επίσης το πού καταλήγει η ενέργεια που χρησιμοποιούμε στον αέρα αλλά και στο νερό, δηλαδή μόλυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναδούμε το θέμα της ε, περιβαλλοντολογικής μας πολιτικής και της ρήπανσης η οποία λαμβάνεται υπόψη με τελείως λανθασμένο τρόπο, ιδιαίτερα όταν κοιτάξουμε την ε, διατροφική αλυσίδα. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο και να μην την απορρίπτουμε με αυτόν τον τρόπο στο έδαφος, στο νερό, κάτι που φυσικά είναι σαν να την ε, αφήνουμε ελεύθερη στα είδη διατροφής που παράγουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το πρόβλημα αυτό με παροπίδες. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους κύκλους παραγωγής κατανάλωσης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για το περιβάλλον και για τη φύση, η φύση συμπεριλαμβάνει δάση, συμπεριλαμβάνει ε, γεωργία και συμπεριλαμβάνει και εμάς. Η στάση μας λοιπόν είναι καθοριστική. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πόλσον. Ο κύριος Χάουσλινγκ, εξ των Πρασίνων. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Κύριε Πρόντι, θα ήθελα και εγώ να σας χαιρετήσω εξ ονόμα της ομάδας μου. Μιλήσατε για την ε, διεθνή ατζέντα. Είναι κάτι που πολύ λίγα πράγματα συμπεριλαμβάνει. Αναφερθήκατε στις επιφάνειες, αναφερθήκατε στη Λατινική Αμερική, και εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν κάποιοι διεθνείς κανόνες. Αλλιώς θα δημιουργηθούν τεράστιες διεθνείς συγκρούσεις. Σήμερα μιλούμε για 6 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία βρίσκονται εγκαταλελειμμένα και υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Χρειάζονται διεθνείς κανόνες. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, γιατί δεν συμφωνώ μαζί σας, είναι αυτή η εντατική εκμετάλλευση της γης. Μιλήσατε για μια αύξηση της παραγωγής της τάξης του 50%. Μα δεν είναι δυνατόν. Με την αλλαγή του κλίματος, οι επιφάνειες τις οποίες μπορούμε να καλλιεργήσουμε θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Η διατροφή, η φτώχεια, δύο αλληλένδετα φαινόμενα. Η πείνα στον κόσμο και βεβαίως η κατανομή των πρώτων υλών και των γεωργικών προϊόντων. Εμείς μπορούμε βεβαίως και έχουμε πολλέ περισσότερες δυνατότητες ο αναπτυγμένος ε, κόσμος. Αλλά τι γίνεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τι γίνεται με τη Λατινική Αμερική και τη βιώσιμη ανάπτυξη η ζήτηση. Μιλήσαμε για το θέμα της σόγιας. Βεβαίως και διαφωνούμε. Και οι επιπτώσεις μιας τέτοιας πολιτικής, όπως ξέρετε, στις εθνικές αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών είναι τεράστιες. Δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε με το φαινόμενο της ε, σπατάλης. 13% 30% των ε, γεωργικών προϊόντων και των που παράγονται στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν χρησιμοποιούνται και όπως ξέρετε αυτό το φαινόμενο διαρκώς αυξάνεται. Η επισητιστική βοήθεια, η βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μια μορφή η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση βιώσιμη. Δεν του βοηθάμε να αναπτύξουν τι δικέ του δυνατότητε. Αυτό δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια βιώσιμη ανάπτυξη την οποία θέλουμε να κάνουμε σαν μοντέλο. Ο γεωργός χρειάζεται, όπως ξέρετε, ασφάλεια και μακροπρόθεσμες προοπτικές για την παραγωγή τους. Δεν μπορούμε να πάρουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα και από τη μία μέρα στην άλλη να αντιστρέψουμε τις ε, τάσεις. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο ολοκληρωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για τις επιφάνειες γης, μην ξεχνάτε ότι στον κόσμο θα πρέπει σύντομα να θρέψουμε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή είναι η προοπτική μας. Πώς τη μετράμε και πώς την ενσωματώνουμε. Και γι' αυτό και μίλησα και για την παγκόσμια agenda και γι' αυτό και, ε, και γι' αυτό και μίλησα και για την κερδοσκοπία. Βεβαίως και υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού, υψηλές τιμές, κερδοσκοπία που οδηγήσει αυτά τα φαινόμενα. Και επαναλαμβάνω, για τη ρύθμιση όλων αυτών χρειαζόμαστε διεθνείς κανόνες. Χρειαζόμαστε μια δυνατή πολιτική και στο θέμα του περιβάλλοντος και στην μεγαλύτερη απειλή ε, για τον πλατηνίτη μας που είναι η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε τις ε, δραματικές της συνέπειες στην Αφρική. E Ευχαριστώ Μάρτιν και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρόντι για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για τις ε, ερωτήσεις των συντονιστών όλων των ομάδων και στη συνέχεια θα παρέμβουν οι υπόλοιποι. Παρακαλώ καθηγητά, ξέρω ότι πρέπει να είμαι πολύ σύντομος, λακωνικότατος θα είμαι. Έχουμε μία οικογένεια ερωτήσεων οι οποίες θέτουν το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κερδοσκοπίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και σαφείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε διευκρίνιστες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς καμία υπερεθνική αρχή η οποία να έχει τη δύναμη, την εξουσία να επιβάλλει κανόνες, το πρόβλημα της ε, κερδοσκοπίας δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιλωθεί. Και γιατί αυτό. Διότι η θεμελιώδης αρχή είναι η πολιτική αυτή να τηρείται από όλους ή τουλάχιστον να την τηρεί μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε εμείς στο G20 παρουσιάζονται κάποιες λύσεις οι οποίες είναι εκ δαμέτρου αντίθετες ε, μεταξύ των για κάθε χώρα και υπάρχουν για παράδειγμα κάποιες γαλλικές προτάσεις οι οποίες κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ λογικές. Εάν όμως αυτές οι προτάσεις δεν υιοθετηθούν από όλους δεν έχουν καμία αξία. Με άλλα λόγια υπάρχει μια αντίφαση παγκόσμιες αγορές και έλεγχοι που θέλουν τα κράτη-μέλη να κρατήσουν στα χέρια τους ε, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους εθνικούς φορείς, τους εθνικούς παραγωγούς. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντίποση, με πάσα ειλικρίνεια πρέπει να σας πω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μία αποτελεσματική λύση. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες τεχνικές προσαρμογές, κάποιες τεχνικές διορθώσεις, αλλά δεν έχουμε λύση. Δείτε λίγο τι συνέβη αμέσως μετά την κρίση. Για πέντε ε, μήνες έπρεπε να ε, κάνουμε αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Ωραιότατες προτάσεις, όλοι με ωραίες ιδέες και τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς κάποιες προσαρμογές ενδιαφέρουσες οι οποίες ε, βελτιώνουν πτυχές διαφάνειας και επιμόρφωσης αλλά από πλευράς κερδοσκοπίας, από πλευράς ε, των hedge και των παραγόγων που απλώς όνομα άλλαξαν αλλά η κερδοσκοπία, η χρηματοπιστωτική πτυχή η οποία είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα είναι τεράστια. Έχουμε επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα, δεν θα πω στα προηγούμενα, αλλά στα επίπεδα τουλάχιστον που είχαμε λίγο πριν από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή ότι ή θα επιδείξουμε σθένους και θα δώσουμε την εξουσία σε κάποια υπερεθνική αρχή ή τουλάχιστον να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ των μεγάλων χωρών επί των θεμάτων για λύσεις ή απλώς θα το συζητάμε για να σώσουμε τις ψυχές μας. Η λύση δεν είναι κοντά δυστυχώς, είναι μια γενικόλογη συζήτηση διότι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο από πολιτική σκοπιά είναι σαφές. Η ίδια συζήτηση είναι η μεταρρύθμιση των διεθνών νομισματικών συστημάτων. Υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες ε, έχουν το κέρδος στο εξωσύστημα είναι αυτός ο οποίος ε, έχει την τον τελευταίο λόγο για το νομισματικό σύστημα, δεν ενδιαφέρεται να νιώσει το διεθνέ νομισματικό σύστημα. Χώρε όπω η Ινδία και η Κίνα επίση δεν ενδιαφέρονται, διότι σε μερικά χρόνια θα έχουν πολύ περισσότερα πόσα έχουν αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή είναι όλα ρευστά και επαναλαμβάνω, ή θα αλλάξει η παγκόσμια διακυβέρνηση ή μην περιμένετε και πολλά από αποτελέσματα. Συγγνώμη που είμαι τόσο ειλικρινής και τόσο σαφής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής ενώπιόν σας. Κάποιες άλλες ερωτήσεις αφορούσαν το θέμα της ε, μη βιωσιμότητας του παρόντος μοντέλου ανάπτυξης. Συμφωνώ απολύτως. Ε, άλλωστε, σα το είπα και εγώ προηγουμένως, το θέμα της κατασπατάλησης ε, είτε πρόκειται για σπατάλες που οφείλονται σε τεχνικές ε, ε, πτυχές, ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αλυσίδα, είτε σπατάλες που κάνει ο ίδιος ο καταναλωτές, δεν πάβουν να είναι πολύ σημαντικές και αυτό το μοντέλο κατανάλωσης πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω πώς και πόσο, ίσως ένα γεωργικό πρόγραμμα, δεν ξέρω αν μπορεί ένα δικό μας ε, γεωργικό πρόγραμμα να βοηθήσει να αλλάξει αυτή η αλλαγή που είναι αλλαγή νοοτροπίας. Δεν αρκεί να αλλάξει το σύστημα των τιμών για να αλλάξουν τα πάντα. Είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα. Επομένως θα πρέπει να ε, κρυούμε τον κόδωνα του κινδύνου συνεχώς, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και τι όρια έχει η δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε. Εδώ τώρα τίθεται το εξή και θα ήθελα να είμαι σαφής. Παράγουμε συνεχώς, ε, είπε και η κυρία Πόλσον ότι ε, παράγουμε με μεγάλη ένταση και δεν έχει έρθει αυτή η στιγμή που θα βάλουμε ένα φρένο. Η αλλαγή στον τρόπο διατροφής είναι αναπόφευκτη. Είναι σχεδόν φυσικό δικαίωμά μας. Σας καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε κυρία Πόλσον, αλλά από την άλλη υπάρχει και η δυσκολία σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένω ιδιαίτερα στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης. Και εδώ θα ήθελα, επιτρέψτε μου να σας δώσω και μια συμβουλή, παρόλο που ίσως δεν ε, είναι και απολύτως αρμοδιότητές μου. Αλλά στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να υποστηρίξουμε με ιδιαίτερο σθένος να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία έρευνας στο γεωργικό τομέα. Η έρευνα ε, ακολουθεί τάσεις, μεγάλες οικογένειες έρευνας. Η γεωργική έρευνα έχει τεθεί στο περιθώριο. Υπάρχουν όμως χώροι οι οποίοι είναι απόλυτα συμβατοί με όλες τις ιδεολογίες που έχουμε για τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς, οι οποίες παραμελήθηκαν διότι δεν επενδύουμε πλέον στη γεωργία. Τα στοιχεία για τη μείωση στην έρευνα για τη γεωργία ε, είναι ε, εντυπωσιακή. Τα στατιστικά στοιχεία είναι απίστευτα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας κάνω μια σύσταση. Τώρα, το land grabbing αυτή η αρπαγή της γης, η επεκτατική πολιτική. Πρόκειται για ένα ε, θέμα το οποίο απορρέει από πολιτικές αποφάσεις που είναι πέραν της γεωργικής πολιτικής. Μία χώρα που έχει, λέει, έχω ένα δις 300 εκατομμύρια πολίτες, ένα δις ε, ε πολίτες, αναφέρομαι στην Ιδία και στην Κίνα. Πολλό δε μάλλον η Κίνα που στα μέσα του αιώνα θα έχει περίπου 1 δισεκατομμύριο 700 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι σαφέ ότι θέτει το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας ως απόλυτη προτεραιότητα και κυρίαρχη ε, πτυχή τη πολιτικής της. Ας ξεχάσουμε τώρα τις μορφές των συμβάσεων. Το να προσπαθήσει λοιπόν να βρει επιπλέον εδάφη, όταν από τις εσωτερικούς τους υπολογισμούς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει επαρκής ε, διατροφική παραγωγή, αποτελεί πολιτική και στρατηγική επιλογή αναπόφευκτη. Γι' αυτό ακριβώ και τίθεται το θέμα τη έρευνα, τη παραγωγικότητα, τη παγκόσμια διακυβέρνηση, τη αλλαγή του τρόπου ανάπτυξη. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Αλλιώς αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, το να χρησιμοποιήσουμε τις κενές εκτάσεις ε, παγκοσμίω είναι πολύ σημαντικό. Τίθεται και το όλο θέμα της χρήσης των υδάτων. Αλλιώς όλες αυτές οι ε, στρεβλώσεις θα είναι αδύνατο να ανακοπούν διότι θα έρχεται η φτωχή κόρα η οποία θα δίνει προς ενοικίαση τις ε, εκτάσεις τους, θα υπάρχει μια χώρα που θα χρειάζεται τρόφιμα και θα είναι διατεθειμένη να πληρώσει πολύ ψηλά ποσά και δεν είναι μόνο η Ινδία και η Κίνα, νομίζω ότι είναι οι χώρες του κόλπου αυτές οι οποίες πρώτες άρχισαν να εφαρμόζουν συγκεκριμένη πολιτική και γιατί φυσικά είναι σαφές ότι οι ίδιοι έχουν προβλήματα νερού και κόστους της γεωργίας που είναι πολύ ψηλό και φυσικά έχουν και στη διάθεσή τους ε, ρευστό αυτή τη στιγμή. Ε, είναι λοιπόν ένα πολύ σαφές ε, πρόβλημα και είναι πολύ κατανοητό ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή λοιπόν η έλλειψη διακυβέρνησης παγκοσμίω πρόβλημα το οποίο ανακύπτει από όλε τι πλευρέ, από όλε τι πτυχέ τη ζωή μα. Και αυτό, κατεμέ με είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο φοβούμε ότι θα το σέρνουμε συνεχώς μαζί μας διότι είναι ε, ε, η σαφής ε, πτυχή που ανακύπτει στη συγκυρία και στην ιστορική στιγμή της αλλαγής εξουσίας. Είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως. Ευχαριστούμε καθηγητά Πρόντι. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις ε, των υπολείπων. Βέβαια οι απαντήσεις σας και τα... είναι τέτοια εμβάθυνση που κάνετε που έχουν ζητήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο. 14 έχω εγγεγραμμένους στον κατάλογο. Θα πρέπει λίγο να προσέξουμε και το χρονοδιάγραμμα γιατί όπως γνωρίζετε στις 11.30 ε, με 12 παρά 20 πρέπει να τελειώσουμε. Ο κύριος Ταραμπέλα και ο Νόμις Άλτον Ντόρφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση. Κύριε Πρόντι, να μπορεί κανείς να ακούει μια τέτοια ομιλία. Όπως και ο Ζακ Δελόρ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, και εσάς, αλλά και ο Ιωσπιζάνη και ο Μισελ Μπαρνιέ, που συμμετέχουν σε ένα think tank αλλά και στα γραπτά του που περιγράφει ακριβώς τους μηχανισμούς που μας περιγράψατε και εσείς, διαπιστώνουμε ότι αυτά που μας είπατε, ότι πρώτον, αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, πάμε προς ε, πολύ σημαντικές ελλείψεις, αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και έλλειψη προϊόντων. Όπως λοιπόν πολύ σωστά μας είπατε, οι πολιτικές δεν μπορεί να συνεχίσουν. Ερωτώ λοιπόν, μήπως πρέπει να βγει η γεωργία από τους μηχανισμούς του διεθνούς εμπορίου. Η Τόχα σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο και υπάρχουν οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής που μας ε, υποβάλλουν προτάσεις διμερών σχέσεων εμπορικών που συμπεριλαμβάνουν βεβαίως και τα γεωργικά προϊόντα, κάτι που ενδεχομένως δεν καλύπτουν πάντα όλες τις ανάγκες ε, των πληθυσμών. Μήπως λοιπόν δεν θα πρέπει να βγούμε από αυτές τις διμερείς είτε διεθνείς συμφωνίες για να μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες που να καλύπτουν σε περιφερειακή ε, βάση τις ανάγκες των πληθυσμών, κυρίων των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών. Τώρα, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό της ε, αρπαγής των γεών το G20 που βεβαίως εκπροσωπεί κυρίως αναπτυγμένες χώρες και προωθεί τα δικά του συμφέροντα, δεν μπορεί να βρει λύσεις. Ενδεχομένως ε, ο ΙΕ ή κάποια άλλη δομή, κάποιος άλλος οργανισμός που θα μπορούσε να επιλεφθεί του φαινομένου αυτού και να επηρεάσει ενδεχομένως μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις πολιτικές έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν καταρχήν οι βασικές ανάγκες των πληθυσμών. Η τροφή και βεβαίως το πόσιμο νερό. Πριν προχωρήσουμε στη δημιουργία υποδομών, κυκλοφορίας ή άλλες υποδομές, θεωρώ σαν προτεραιότητες επενδύσεις στον γεωργικό τομέα για τα βασικά γεωργικά προϊόντα, τα απαραίτητα για την ζωή και αυτό σε περιφερειακή κλίμακα. Ευχαριστώ πολύ ο Μισελ Νταντέρ και κατόπιν ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον καθηγητή για την ομιλία του. Έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν δύο διαφορετικά θέματα. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς ε, προβλέψεις. Ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής στο τέλος της χιλιετίας και ήσασταν από τους πρωταγωνιστές ε, των ε, διαβουλεύσεων για τον προϋπολογισμό και τις δημοσιονομικές προβλέψεις. Σήμερα βλέπουμε νέους παρεμβαίνοντες όπως η Κίνα και η Ινδία που δεν ήταν εύκολο να προβλεφθεί η δράση τους. Μπορείτε να μας πείτε γιατί το 2000-2003 η ανάλυση που έγινε ήταν εσφαλμένη όσον αφορά αυτά που συνέβησαν μετά το 2004-2005 και που μας οδήγησε στην κρίση στον τομέα των ειδών διατροφής. Δεύτερη ερώτηση. Έχουμε ένα επιστημικό μοντέλο στην Ευρώπη που είναι εξαιρετικά περίπλοκο με κανόνες που βεβαίως ε, δίνουν μια ασφάλεια στον καταναλωτή, πολύ μεγάλη ασφάλεια. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των πληθυσμών της γης με μοντέλα τα οποία να μπορεί να εξάγονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, εκτός Ευρώπης δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ, ο Μισελ Ντόρφμαν και κατόπιν ο Ζεζέ Μποβέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε καθηγητά για τα όσα μας είπατε, τα οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αναφερθήκατε στην ε, απώλεια εκτάσεων που έχουμε σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο συχνά δεν αναφέρεται στον κατάλογο των εταίων και υπάρχει και η εγκατέλειψη ε, καλλιέργειας σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι απλώς προσοδοφόρα η καλλιέργεια. Κάποιος ε, γεωργός δηλαδή φεύγει γιατί δεν έχει οικονομικά ωφέλη από την καλλιέργεια. Στην ε, Ιταλία καταλήφθηκαν εκατοντάδες ε, χιλιάδες εκτάσεις διότι δεν μένει πλέον κανείς στις Άλπεις, στα Απένινα και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Αυτό που διαρωτώμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι αν η γεωργική πολιτική που κάνουμε οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση αν μπορέσουμε να ανακόψουμε δηλαδή το φαινόμενο αυτό που οφείλεται και σε θέμα γενεάς. Πολλές φορές εγκαταλείπουμε τις εκτάσεις ε, λόγω γενεών. Οι παλιοί συνεχίζουν και όταν έρχονται οι νέοι δεν θέλουν πλέον να καλλιεργήσουν μια έκταση και φεύγουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολύ συχνά δεν αναφέρεται, δεν αναφέρεται ποτέ μάλλον και ποτέ δεν ε, επισημαίνεται. Νομίζω ότι όμως τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή ως προς την ανάγκη χρήσης της γης θα πρέπει να κάνουμε και τη συγκεκριμένη συζήτηση, να αναφέρουμε και αυτή την πτυχή. Είπατε κι εσείς ότι θα υπάρξει σίγουρα αύξηση των ε, τιμών των γεωργικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, δεν ξέρω και αν η κοινή γεωργική πολιτική με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή στον πρώτο πυλώνα είναι και η πραγματική την απάντηση, διότι η αύξηση των τιμών ουσιαστικά πρημοδοτεί αυτόν που μπορεί να παράγει περισσότερο στις πιο ευνοημένες περιοχές της Επίρου μας, οι οποίοι θα είναι και αυτοί που θα έχουν τις υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα. Και να αναφερθώ στην πολύ σωστή σας παρατήρηση για την τεχνολογική ανάπτυξη. Δυστυχώς εγώ έχω την εντύπωση ότι στη γεωργία σε αντίθεση με όλους σχεδόν τους υπόλοιπους τομές, ε, συχνά αποφεύγουμε την τεχνική. Είμαστε κατά της τεχνικής. Σήμερα θεωρούμε ότι είμαι σύγχρονη ε, και εμείς επιστρέφουμε στους καιρούς των προγόνων μας. Κανείς άλλος δεν το κάνει. Όλοι οι άλλοι βιομηχανικοί τομείς ε, δεν παράγουν προϊόντα με τον τρόπο που, θα το, που το έκανε η πρόγραμμή μας. Ενώ στη Γεωργία δυστυχώς συχνά είναι έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν, ο Ζωζέ Μποβέ τώρα, ο Αντιπρόεδρος και κατόπιν ο κύριο Νικολέσκου. Κύριε Πρόντι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εκτίμησα τα όσα είπατε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, χωρίς να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου. Δύο-τρεις παρατηρήσεις λοιπόν. Πριν από λίγο μας μιλήσατε για το ζήτημα της διατροφής, ότι θα πρέπει να ταΐσουμε τον πλανήτη και είπατε έπειτα ότι πρέπει να υπάρχουν και παγκόσμιες ρυθμίσεις για τις χώρες. Δεν πιστεύετε ότι το ζήτημα αυτό δεν θα πρέπει να το καθορίσει ούτε το G8 ούτε το G20 αλλά τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι θεμελιώδες σήμερα, αν πραγματικά θέλουμε να ρυθμίσουμε παγκοσμίω την κατάσταση, να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα στη διατροφή, το οποίο όμως δεν αρκεί από μόνο του. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σε διεθνές επίπεδο όλο και περισσότερα άτομα και ο κύριος Δεγκούτερα, ο εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών, λένε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην διατροφική κυριαρχία προκειμένου οι χώρες μεμονωμένα να μπορούν να προστατευθούν από τις μεγάλες πολυεθνικές που πολλές φορές έχουν ε, τάσεις ε, ε, ιδιαίτερα αρπακτικές. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν τα απαραίτητα μέσα, ακόμα και τεχνικά μέσα, προκειμένου μια τέτοια πολιτική να εφαρμοστεί. Πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί η κατάσταση στα πλαίσια των Εθνών να αναγνωριστεί για κάθε χώρα το δικαίωμά τη στη διατροφική αυτή κυριαρχία. Δεύτερον, όσον αφορά την παραγωγικότητα, συμφωνώ μαζί σα, υπάρχει πρόβλημα παραγωγικότητα. Το θέμα όμω αυτό δεν τίθεται ούτε στην Ευρώπη ούτε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει να κάνει κυρίω με τι ε, χώρες του νοτίου ημισφαιρίου όπου πραγματικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από τις δυτικές ε, χώρες, τις χώρες του βορείου ημισφαιρίου. Βλέπουμε ότι στις ε, χώρες αυτές πρέπει να υπάρχει απαραίτητη ανεπτυξιακή βοήθεια προκειμένου οι χώρες αυτές να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όλο το γεωργικό δυναμικό παραγωγής το οποίο έχουν. Και αυτό πάλι στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ρυθμιστεί, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι χώρε αυτέ και να μπορούν να βαρύνουν περισσότερο στο παγκόσμιο προσκήνιο. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα, σαφώ θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο η έρευνα, αλλά για άλλη μια φορά και εδώ θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι η βασική μας ανάγκη είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα στις χώρες της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας και ότι θα πρέπει εκεί πέρα να χρησιμοποιηθούν κάποιες απλές τεχνικές προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή στις περιοχές αυτές του κόσμου. Να λοιπόν τρεις παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω προκειμένου να εμπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και κατά κλείδι να πω ότι ελπίζω ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου σήμερα το απόγευμα θα δείξει το απαραίτητο θάρρος προκειμένου να υπερψηφίσει την έκθεση αυτή που προβλέπει μια θετική εξέλιξη της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο κύριος Νικουλέσκου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Να σε ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που κάνατε σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο σημεία. Όταν μιλάμε για έλλειψη τροφίμων, θεωρούμε ότι αυτό ισχύει για τις φτωχές χώρες. Το φαινόμενο όμως αυτό μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε. Πρόσφατα μία τράπεζα στην Ιαπωνία έκανε μία, ένα κατάλογο των χωρών που πλήττεται περισσότερο από τη διακύμαση των τιμών των τροφίμων. Αναφέρθηκαν στις δαπάνες, στις οικογενειακές που γίνονται για την αγορά τροφίμων και συνδύασαν τις δαπάνες αυτές με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και είδαν ότι υπάρχουν τέσσερις χώρες από τα 27 κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται ιδιαίτερα από την κατάσταση η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Και η Κροατία επίσης και αυτή με τη σειρά της επηρεάζεται από την κατάσταση αυτή. Ο Αμαριτασάν, ένας νομπελίστες είπε ότι ε, δεν θα πρέπει τον επόμενο αιώνα να επηρεαζόμαστε, να θυγόμαστε από την πείνα, από φαινόμενα ένδυας. Δεν νομίζω όμως ότι κάτι τέτοιο θα το αποφύγουμε. Δεν πιστεύετε ότι ε, αν συνεχίσουμε με αυτές τις ε, τάσεις στον προπολογισμό η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι καταδικασμένη. Αναφερθήκατε επίσης στην χρήση των γεών. Η δική μου χώρα έχει μία εξαιρετική δυναμική, δυνα... φοβερέ δυνατότητε όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των γεών. Πάρα πολλέ αρρώσιμε γέε όμω οι οποίε δεν χρησιμοποιούνται. Νομίζω ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να πετυχαίνει μια καλύτερη ισορροπία όσον αφορά τις βοήθειε που δίνονται, τη βοήθεια που δίνεται ανάμεσα στην Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σικυριέσκη τώρα και μετά η Ελίζαμπετ Γέγελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόντι, ήρθατε και μα μιλήσετε σήμερα ενώ συζητάμε το μέλλον τη κοινή γεωργικής πολιτική, καθώ επίση και το μελλοντικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταπληκτική σύμπτωση λοιπόν αυτή όπου βλέπουμε έναν καθηγητή πρώην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα λέει πράγματι ιδιαίτερα θαραλέα. Κύριε καθηγητή λοιπόν, θα μπορούσατε να επαναλάβετε τα όσα λέτε σήμερα αν ήσασταν εκ νέου πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λέγατε τέτοια πράγματα. Μπορώ να φανταστώ βέβαια την απάντηση που θα δώσετε, γιατί κινούμεθα βέβαια στον χώρο της πολιτικής. Ο λόγος που κάνουμε στην παρατήρηση αυτή είναι ότι συνειδητοποιώ ότι δεν έχουμε πλέον όραμα στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που γίνεται είναι θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό κατά 0,1%. Ενώ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όταν φεύγατε εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση που γινόταν τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση του προπολογισμού ήταν της τάξης του 1,24%. Η παρέμβασή σας πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Το μόνο το οποίο έλειπε ενδεχομένω ήταν το να εξετάσουμε λίγο περισσότερο τη σχέση παραγωγικότητας και εισοδήματος. Μιλάμε για ανθρώπου, για πληθυσμού οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά και το βιωτικό του επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλε επαγγελματικέ ομάδε. Έχουμε ξεπεράσει πια την περίοδο των χαμηλών τιμών στα τρόφιμα. Και πολλέ φορέ όταν οι τιμέ είναι πάρα πολύ χαμηλέ δεν σεβόμαστε τελικά την αξία των τροφίμων. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει η νοοτροπία κυρίως των πλουσίων κρατών όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια και τα δημόσια αγαθά. Επίσης δεν αναφερθήκατε πολύ στην σχέση τροφίμων και υγείας. Οι δύο αυτές έννοιες είναι σαφώς αλληλένδετες, πιστεύω πρέπει σιγά σιγά να κινηθούμε από μια κοινή γεωργική πολιτική προς μια παγκόσμια στρατηγική ευσυτισμού όλου του πλανήτη. Και έρχομαι στα λόγια σας τώρα όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την παγκόσμια αυτή governance. Δεν ξέρω αν το ζήτημα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει το G8, το G20 ή τη συνελεύση των ΗΕ. Πάντως χρειαζόμαστε σαφώς μια παγκόσμια ρύθμιση στη γεωργία. Ως απόρρια της παγκόσμιας κρίσης έχουμε δημιουργήσει κάποια σώματα ρυθμιστικά για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε χρηματοδοτήσει με πάρα πολύ υψηλά ποσά τις αγορές αυτές, τόσο στην Ευρώπη όσο, όσο παγκοσμίω. Για ποιο λόγο δεν κάνουμε κάτι ανάλογο και με τον γεωργικό αγροτικό τομέα. Ξέρετε ότι είναι ένα τομέα ο οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τη ρύθμιση δύο-τριών παραγόντων, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί εξωτερικοί παράγοντε που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα, όπω οι κλιματικέ αλλαγέ. Επομένω, α μην δείχνουμε πλέον δηλία, α ρυθμίσουμε θαραλέα παγκοσμίω και τον αγροτικό τομέα. Και τέλο, όντω χρειαζόμαστε περισσότερη επιστημονική έρευνα. Πολλές συζητήσει γίνονται για την καινοτομία, για καινοτόμο τεχνολογία την οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά. Αναφερόμαστε σε επιστημονική έρευνα όσον αφορά τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Τέλος να σας πω ότι εύχομαι η προσέγγιση την οποία πρεσβεύεται να δίνει πραγματικά η παγκόσμια προσέγγιση. Ε, ε, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, ε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη με τον Επίτροπο τότε Φίσλερ ήταν αυτοί οι οποίοι ηγήθηκαν της μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής η κυρία Γέγκλε και μετά η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε καθηγητά. Μας παρουσιάσετε πολλές σκέψεις, πολλά πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν και εμάς σε σκέψη και περισυλλογή. Ο καθένας ενδεχομένως μόνος του και κατόπιν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και εδώ στην Επιτροπή. Κύριε Πρόντι, Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, στο γύρο της Ντόχα. Ένας αδύναμος γύρος θα έλεγα, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά προς το παρόν. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην σειρά διμερών συμφωνιών που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η θέση σας για αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις συμφωνίες οι οποίες είναι περιορισμένες, λύνουν ή δεν λύνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα αγνοώντας ε, το συνολικό πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, αυτού του είδους οι εμπορικές συναλλαγές χάνουν τον γενικό σκοπό της πολιτικής μας. Ευχαριστώ πολύ. Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον καθηγητή Πρόντι. Αναφερθήκατε στην ομιλία σας δύο φορές στο ηθικό μας καθήκον. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει πιο συχνά να το χρησιμοποιούμε σαν έννοια. Έχουμε αρχίσει να το χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το τραπεζικό σύστημα, διοντολογία και ηθική. Θα έπρεπε ίσως να το χρησιμοποιούμε και για την πρόσβαση στην τροφή. Να μιλάμε δηλαδή για ηθική, για δεοντολογία και σωστή ρύθμιση αυτού του τομέα. Μιλήσατε για την ανάπτυξη. Κύριε Πρόντι, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όσον αφορά παραδείγματο χάρη την έρευνα και τη χρηματοδότησή της. Υπάρχουν χώρες που έχουν σταματήσει την δημόσια στήριξη αυτής της έρευνας. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κρατική δημόσια χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν αυτή την έρευνα. Και χαιρετίζω ιδιαίτερα το ότι έχει αρχίσει να μας απασχολεί το θέμα αυτό. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι οι πλούσιες χώρες δεν πρόκειται να πεινάσουν. Αυτό είναι γεγονός. Αν κάποιος όμως βρίσκεται μεταξύ αυτών που πεινούν και πολλοί σήμερα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ε, βοηθήσουμε η πρόσβαση στα τρόφιμα, στην τροφή και στο πόσιμο νερό είναι κάτι που σαφώς θα πρέπει να το δούμε με έναν ισορροπημένο τρόπο. Το δικαίωμα στην επιστημιστική ασφάλεια, στην παραγωγή τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να το δούμε, το φαινόμενο αυτό. Όσον αφορά τώρα το τρίτο θέμα που θα ήθελα να θίξω, που είναι η αρπαγή της γης, μεγάλες επιφάνειας γης στην Αφρική, βρίσκονται σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο ολοκληρωμένα. Δηλαδή αν χρειάζεται κάποιος αυτές τις επιφάνειες για την παραγωγή τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο να το δούμε πολύ πιο γενικά και ολοκληρωμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόντι, αναφερθήκατε στις χώρες αυτές οι οποίες έχουν αρχίσει την εξαγωγή ε, ειδών διατροφής. Και σας άκουσα να επικρίνετε αυτό το ε, φαινόμενο στα πλαίσια των συμφωνιών και της πολιτικής του ΠΟΕ. Όμως οι διάφορες χώρες έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική έτσι ώστε βλέπουμε ότι πολλές φορές χάνεται ο συνολικός στόχος. Δημιουργούμε δηλαδή αποθέματα την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικές στάσεις βάσει αυτών των αποθεμάτων. Ακούγοντας αυτά που είπαμε εδώ, θα ήθελα κι εγώ να πω ότι δεν αναφερθήκατε σε ένα πάρα πολύ προφανές θέμα για μένα. Τις λύσεις. Τις λύσεις. Πρέπει να παράγουμε βεβαίως τροφή. Και το θέμα είναι τι κάνουμε με τις νέες τεχνολογίες που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας, όπως παραδείγματος χάρη τους τροποποιημένους γενετικά οργανισμούς. Δεν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο Ζωζέ Μποβέ κάθεται λίγα μέτρα δίπλα σας και αυτό σας απέτρεψε. Μη φοβάστε όμως, δεν είναι τόσο δυνατός και τόσο ψηλός. Μπορείτε να αναφερθείτε στο θέμα αυτό. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας άλλος πράσινος μίλησε για τα θέματα αυτά χωρίς όμως να αναφέρει λύσεις. Και είχε δίκιο. Χρειαζόμαστε λύσεις. Πολλά από τα τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, που δεν χρησιμοποιούμε, πολλά από τα αποθέματα δεν ρυθμίζονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου όμως θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Αφού βεβαίως προηγουμένως τα προϊόντα αυτά έχουν ε, σημανθεί. Θα ήθελα να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όπως παραδείγματος χάρη παραγωγή σόγιας ή τα ψάρια τα οποία τα ξαναπετάμε στη θάλασσα. όσον αφορά τις ζωοτροφές, όσον αφορά τα θηλαστικά που ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις τρέφονται με τροφές οι οποίες δεν θα έπρεπε. Δηλαδή βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνονται κρέατα στις τροφές τους. Θα ήθελα... Και τώρα ο κύριος Γιάρ και μετά ο κύριος Πρόντι που θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Πρόντι. Ο κύριος Γιάρ. Πολλές ερωτήσεις ήθελα να κάνω, τις έκαναν όμως οι συνάδελφοι πριν από μένα. Κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα γίνει αντικείμενο ερώτησης είναι οι διακυμάνσεις των τιμών, έντονες διακυμάνσεις. Επίσης, οι πολιτικοί που ασχολούνται με το θέμα της γεωργίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αντικείμενα κριτικής όσον αφορά τις επιδοτήσεις ε, στις εξαγωγές και τις επιπτώσεις βεβαίως στις τιμές. Εγώ σήμερα είπα βεβαίως και το ξαναλέω ότι το πλεονέκτημα της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις. Και οι τιμές βεβαίως σήμερα αυξάνονται. Θα συνεχίσουν να αυξάνονται άσχετα από τις διακυμάνσεις τις οποίες δεν θέλουμε να υπάρχουν. Η ερώτηση μου λοιπόν ίσως σας φανεί λίγο αφελής, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Θα πρέπει οι τιμές αυτές που αυξάνονται να αποτελέσουν κίνητρο για καλύτερη και περισσότερη παραγωγή. Θα μπορέσουν αυτές οι αυξημένες τιμές να χρησιμοποιηθούν και να είναι χρήσιμες και ωφέλιμες και για τους αγρότες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το επιληφθούν οι πολιτικοί. Τι κάνουμε με τις εξαγωγές, τι κάνουμε με την αναπτυξιακή μας πολιτική. Αυτό είναι κάτι που σαφώς, όπως βλέπετε, δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας σε σχέση με την πολιτική που αποφασίζουμε σε περιφερειακό επίπεδο και σε σχέση με την ε, Γεωργία. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ρωμάνο. Ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για ένα πρόβλημα το οποίο συμπληρώνει αυτά τα οποία συζητήσαμε μέχρι τούδε και ιδίως το πρόβλημα της προσαρμογής της αλλαγές του κλίματος και στην προσαρμογή που πρέπει να κάνουμε στα εδάφη ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει το έδαφος να μπορεί να υποστεί κατάλληλη μετατροπή ώστε να διατηρεί το νερό ε, και να μην έχουμε υποχώρηση των εδαφών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το συζητήσει η Επιτροπή Γεωργίας, διότι νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέργειες τις οποίες θα πρέπει να ε, λαμβάνουμε υπόψη στο σημείο αυτό. Να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στα εδάφη και τα κατάλληλα μέσα για να μετρήσουμε κατά πόσον δίνεται ιδέουσα προσοχή στο έδαφος. Ακόμα και οι δορυφορικές δομές μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μια εικόνα της υγείας των εδαφών και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το έδαφος να παραμείνει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την πρωτογενή του χρήση που είναι η παραγωγή τροφίμων. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ε, το γεγονός ότι πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε και την απερίμωση. Πέρα από την αρπαγή της γης, του land grabbing, υπάρχει και ένα desert grabbing. Θα πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πτυχή, διότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικότερα αίτια Ε, τα οποία οδηγούν ε, τους ε, καλλιεργητές, επειδή ακριβώς πεινούν, να αναζητήσουν διέξοδο αλλού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και τις κατάλληλες δομές ευρωπαϊκά για να διαχειριστούμε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μία τελευταία αμνία στο εξή. Στην Ιταλία έχουμε 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτάσεων τα οποία είναι μολυσμένα. Θα μπορούσε να γίνει κάποιο πρόγραμμα εξυγίανση το οποίο θα μπορούσε να βασιστεί και σε ενεργειακές ε, πολιτικές ώστε βαθμιδών τα εδάφια αυτά να επανέλθουν στην πρωταρχική τους χρήση που είναι η παραγωγή διατροφικών προϊόντων. Ευχαριστούμε τον κύριο Βιτόριο Πρόντι. Ο κύριος Βατσεβόσκι τώρα και κατόπιν Μόρβη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από 7 χρόνια θυμόμαστε πολύ καλά ότι εγκαταλείψατε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα 1,24% του ΑΕΠ όσον αφορά το προπολογισμό. Όντως τότε χρειάστηκε να μειώσετε το ποσοστό αυτό στο 1%. Ενδεχομένω να έχει πειραστεί όμω και η πιστική ασφάλεια εξαιτία αυτού, γιατί θα ήταν καλό να είχαμε περισσότερα χρήματα. Τώρα στην κοινή γεωργική πολιτική έχουμε δύο ομάδε πολιτικών. Αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική και αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να παραμείνει στη ίδια Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες ή μάλλον αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτα αν δεν αυξήσουμε τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι τέτοια ώστε να αποκρίνεται πραγματικά στις νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το 2004 το 2007 μάλλον, πριν την επισητιστική κρίση, πριν αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων, προτού προκύψουν όλες αυτές οι νέες προκλήσεις, προτού ξεκινήσουν ε, οι δραματικές αυτές προβλέψεις που λένε ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα τρόφιμα, να διπλασιαστούν, να αυξηθούν κατά 50-70%. Την εποχή εκείνη μιλούσαμε απλώς για έναν προπολογισμό που νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε και να μειώσουμε, ότι είχαμε την πολυτέλεια να το, μειώσουμε. το Τώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο προπολογισμό. Να αναφερθώ τώρα και στο ζήτημα της αγρανάπαυσης, της εγκατάλειψης κάποιων γεών. Στην Ιταλία, κύριε Πρόντι, ένας γεωργός παίρνει 300 ευρώ ένα εκτάριο γης. Τι γίνεται όμως με τις νέες χώρες όπου τα χρήματα αυτά είναι μόνο 100 ευρώ. Το σύστημα της αγρανάπαυσης στις χώρες αυτές προχωρά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν νομίζω θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα, να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη εξορρόπηση πληρωμών και επιδοτήσεων ανάμεσα σε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά νομίζω ότι θα καταστραφεί η Γεωργία αν δεν έχουμε ένα ισορροπημένο μοντέλο. Κύριε Πρόντι, σα ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά για το θαραλέο προπολογισμό που είχατε προτείνει στην παλαιότερη θέση που είχατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βατσεβόσκη. Μόρβεϊ, η κυρία Μόρβεϊ και μετά ο, Σέρτζιο Σιλβέστρης. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλεγμένοι όλοι πολιτικοί που εκπροσωπούμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ο λόγος που τα λέω όλα αυτά κύριε Πρόντι είναι ότι ε, δεν θέλω να φύγετε από την αίθουσα αυτή, να επιστρέψετε στην χώρα σας πιστεύοντας ότι ε, οι λαοί της Ευρώπης συμφωνούν με την ιδέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Υπάρχουν εκατομμύρια στην Ευρώπη που πιστεύουν ότι ε, η παγκόσμια διακυβέρνηση, η ιδέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι απαράδεκτη και τρομακτική. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Υπάρχουν εκατομμύρια πολιτών που πιστεύουν ότι είναι μια πολύ κακή ιδέα να πάρουμε όλο και περισσότερη εξουσία από τους ανθρώπους και να δημιουργηθεί ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους πολίτες τους λαούς και τους ηθήνοντες που χαράσουν πολιτική. Να αυξηθεί μάλιστα το χάσμα αυτό, μεταφέροντας όλο και περισσότερο την εξουσία λήψης αποφάσεων από τον ίδιο το λαό, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καν εκλεγεί, δεν υπόλογοι σε κανέναν, δεν λογοδοτούν, είναι απλώς γραφειοκράτες, οι οποίοι εργάζονται με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου διαφανής. Να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Πρόντι, αν εσείς και το think tank του οποίου υγείστε έχετε σκεφτεί μία εναλλακτική λύση, μία αντίθετη λύση, να δώσετε πίσω στις κοινότητες, πίσω στους πολίτες και στους λαούς την εξουσία αυτή, να παίρνουν αυτοί αποφάσεις για τον εαυτό τους. Και συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος που συζητάμε, της, του διατροφικού ζητήματος αντί να παγκοσμιοποιηθούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και να συγκεντρωθεί εξουσία σε λίγους, μήπως θα πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο, δηλαδή αποκέντρωση, επιστροφή της εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες και στους λαούς. Ακούσαμε και την ιδέα της διατροφικής κυριαρχίας. Ως προς αυτό γίνονται σπουδαία πράγματα, κυρίως στα Έθνη, όπου θέλουμε πραγματικά η διατροφική κυριαρχία να γίνει ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκαμε επίση στο ζήτημα του ελέγχου των γεών όσον αφορά τη διατροφική κυριαρχία. Και κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και οι τοπικέ κοινωνίε θα πρέπει να είναι σε θέση οι ίδιε να αποφασίζουν τι θέλουν να παράγουν, πώ θα το παράγουν, πώ θα το πουλάνε. Και θα πρέπει και οι καταναλωτέ, οι μεμονωμένοι πολίτε, να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υγιή τρόφιμα, όχι σε οποιαδήποτε τρόφιμα, σε υγιή τρόφιμα και καταλαβαίνετε ότι γη είναι τα τρόφιμα αυτά τα οποία παράγονται τοπικά, αυτά τα οποία είναι φρέσκα. Κύριε Πρόντι, λοιπόν, μήπως θα ήταν μια καλύτερη ιδέα να επιστραφεί η εξουσία η δυνατότητα λήψης απόφασης στους ίδιου τους πολίτες, να αποφασίσουν αυτοί πώς θα παράγουν, τι θα παράγουν και πώς θα καταναλώνουν τα τρόφιμα αυτά. Μήπως θα πρέπει να αποφύγουμε την μη δημοκρατική λύση της παγκόσμιας διακυβέρνηση. Ευχαριστούμε κυρία Μορβέη. Ο Σέργιο Σιλβέστρη είναι αυτό που θα κλείσει το κύκλο ερωτήσεων τη Επιτροπή μα. Σέργιο, έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πρόεδρε Ντεκάστρο, ευχαριστώ και τον πρόεδρο Πρόντι για την παρουσία του εδώ και για την προσοχή που δίνει σε θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά για μα. Μα τα παρουσίασε άλλωστε σήμερα και πολύ επίκαιρα διότι με μεγάλη ικανοποίηση αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά στα πρόθυρα πολύ σημαντικών θεμάτων που θα ε, απασχολήσουν την Επιτροπή μας. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε λίγο πράγματα ε, παραπάνω και εσείς μας δώσετε σίγουρα τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ γι' αυτό. Θέσατε το θέμα των γεών το καθορίσατε και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ε, πρόκειται για μία από τις τρευλώσεις που δεν θα μπορέσουμε να ανακόψουμε. Ε, θα έχουμε αρπαγή γης ε, σε εκτάσεις από χώρες οι οποίες είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Υπενθυμίσε επίσης ο Βιτόριο Πρόντι και το γεγονός ότι η εγκατάλειψη των γεών δημιουργεί πολύ σημαντικές δυσκολίες. Εγώ στο θέμα αυτών λοιπόν των ε, εκτάσεων προς εκμετάλλευση θα ήθελα να θέσω και ένα ε, πρόβλημα το οποίο βιώνουμε στην ε, Ιταλία αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές πλέον είναι εκμεταλλεύσιμες με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργία. Τους τελευταίους μήνες διαπιστώνουμε ότι πολλές γεωργικές επιχειρήσεις πτωχεύουν λόγω δυσκολιών και αγοράζονται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γεννηθεί λίγες πριν, ε, μέρες ε, πριν και δεν έχουν καμία ε, σχέση με τη γεωργία. Σε περιοχές που πολύ δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε. Ξέρετε ότι ένας μικρός δήμος, για παράδειγμα, τον οποίο πολύ δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε και δεν μπορεί να ελέγξει τι γίνεται, όπως το Ταραντίνο, για παράδειγμα, ή σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, και οι δομές είναι μικρές. Αυτό λοιπόν που ελοχεύει ως κίνδυνος είναι ότι πολλές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αποτελούσαν ε, δυνατότητα για να παράγουμε καρπούς θα γίνουν πλέον ε, διαφορετικοί χώροι που θα τυχάνουν άλλες εκμετάλλευσεις που δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργία. Θα ήθελα να θέσω λοιπόν και αυτό τον προβληματισμό στο πρόβλημα των εκτάσεων που θέσατε. Όσον αφορά τώρα την επισητιστική ασφάλεια, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρέπει να, όπως είπατε και εσείς, να προσέξουμε περισσότερο την έρευνα, να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια προοπτική για όλη αυτή τη λογική που μας εκθέσετε. Πέρσι όμως ο πρόεδρος Δεκάστρο στην ε, ημέρα που κάναμε για την ε, κατασπατάληση των τροφίμων ε, έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Στις ανεπτυγμένες χώρες, στις χώρες της Δύσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γεωργικών προϊόντων, το 20%, πετιέται. Από και ξέρετε ότι με αυτό το 20% θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα για το 1 δισεκατομμύριο του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το ε, κατόφλι της ε, ελάχιστης δυνατής σύντησης. Νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα της επιστημιστικής ασφάλειας θα μπορούσαμε να το ε, εξετάσουμε και από την πτυχή αυτή των αποβλήτων. Μία τελευταία παρατήρηση, η σχέση των νέων με τη γεωργία. Νομίζω ότι οι νέοι μπορούν να διαδραματίσουν πολύ ουσιαστικό ρόλο για τη γεωργία. Μπορούμε να έχουμε νέους πόρους, νέες ε, δυνατότητες, ακόμα και διαφορετική νοοτροπία προσέγγισης του συστήματος και του επαγγέλματος του γεωργού. Μέχρι τώρα όμως οι πολιτικές για τους νέους, οι οποίες σχετίζονται μόνο σε μία πρώτη βοήθεια για την ένταξή τους, είναι πολύ ισχνές. Εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ενταχθούν και οι νέοι στη γεωργία, με τη συνοδεία φυσικά και αποτελεσματικών πολιτικών, όπως προτείναμε για παράδειγμα εδώ στην Επιτροπή να υπόστη ρίξουμε την ε, ανασύνθεση συγκεκριμένε επενδύσει. θα αποτελούσε νομίζω μεγάλο πλεονέκτημα για τον τομέα. Πραγματικά σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Πρόντι για την παρουσία σας και για την ε, σημασία των όσων είπατε. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους ε, που πήραν το λόγο σε αυτή την τόσο σημαντική και έκτακτη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Να ευχαριστήσω και σένα αγαπητέ Ρωμάνο, διότι μας έδωσες μια εξαιρετική ευκαιρία ε, μας παρουσίασες μια εσβάθος ανάλυση των πραγμάτων, να αυξάνονται και οι ευθύνε μας από εδώ, όπως υπενθύμησα, αλλά μπόρεσες να δεις και λίγο πώς είναι οι διαφορετικές ευαισθησίες των Ευρωβουλευτών, των διαφόρων πολιτικών ομάδων της Επιτροπής μας. Να σου δώσω λοιπόν το λόγο, όση ώρα θες για να απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, τις πάμπολες ερωτήσεις που σου τέθησαν. Ευχαριστώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω πολύ από το χρόνο σας, διότι θα ήταν απειλή. Αυτή τη συζήτηση πραγματικά την βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και γιατί ποικίλουν οι διάφορες θέσεις, και φυσικά ποικίλουν και οι ευαισθησίες και αυτές τι ευαισθησίες θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη απολύτως. Πρώτος προβληματισμός, το θέμα του διεθνούς εμπορίου. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσε θέσεις. Αφενός ε, θα έλεγα η πιο ενδιαφέρουσα άποψη ήταν ε, αυτή της κυρίας Μορβέη, η οποία μας είπε ότι προσέξτε, εδώ δεν λειτουργεί το μοντέλο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, οπότε ας ξαναδώσουμε την εξουσία σε τοπικό επίπεδο. Θεωρητικά είναι τέλεια αυτή η άποψη. Το θέμα είναι όμως τι σημαίνει από οικονομικής πλευράς η εξουσία να περάσει σε τοπικό επίπεδο. Σημαίνει ότι καταρχάς οι τιμές και το κόστος ε, θα ανέβει κατακόρυφα, διότι γνωρίζετε ότι χωρίς την παγκόσμια συνεισφορά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα λογικό σύστημα και δεν θα έχουμε και διαθεσιμότητα αγαθών. Διότι ακόμα και η διαφορά του μικροκλίματος ε, δεν επιτρέπει να υπάρχει επάρκεια σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον όχι απόλυτη επάρκεια. Θα πρέπει μεν λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις ε, τοπικές ιδιαιτερότητες, να ευνοήσουμε επίσης ε, και την, ε, το τοπικό μάρκετινγκ, την προώθηση προϊόντων σε τοπικό επίπεδο, αλλά το να είμαστε αποκλειστικά και μόνο σε τοπικό επίπεδο σημαίνει ότι θα ανέβουν κατακόρυφα οι τιμές και μάλιστα με, σε τιμές τις οποίες πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο ανέφεραν πολλοί από εσά. Το να αποδεσμευτούμε από τους διεθνείς μηχανισμούς, ε, να είμαστε υπέρ περιφερειακών ή συνολικών συμφωνιών, υπάρχει μια διαβάθμιση. Κάποιοι λένε να προωθήσουμε, να πρημοδοτήσουμε την τοπική αγορά, κάποιοι την περιφερειακή, κάποιοι την παγκόσμια. Ανάλογα με τη λύση που θα επιλέξουμε φυσικά υπάρχουν και διάφορες ε, εκφάνσεις της κατάστασης. Αν και διατηρήσουμε την αγορά σε τοπικό επίπεδο, σαφώς υπάρχουν δυνατότητες πιο ισχυρού κοινωνικού ελέγχου. Αλλά υπάρχουν και πολύ πιο αυξημένες τρευλώσεις των τιμών. Ακόμα και οι διμερείς συμφωνίες, από την ε, εμπειρία μου, ε, διότι φυσικά επειδή δεν υπάρχει και συμφωνία στο γύρο της Δόχας ε, είναι πιο διαδεδομένες είναι πολύ πιο ε, σημαντικές για αυτούς που δεν συμμετέχουν στη διμερή συμφωνία. Ε, πρόκειται δηλαδή για μια δεύτερη επιλογή σε σχέση με το καλύτερο που χρειαζόμαστε. Εδώ όμω επανερχόμαστε στο πρόβλημα που μου θέσετε. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνει τη Γενική Συμφωνία, το G20, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΙΕ. Αυτή τη στιγμή ως έχει κατάσταση νομίζω ότι ήμουν και ιδιαίτερα ειλικρινής και σας είπα ότι πόρο απέχουμε από την ε, δυνατότητα να αναλάβει κάποιος την ευθύνη αυτής της μορφής. Διότι το G20, το οποίο στη θεωρία είναι η δέσμευση, ο συμβιβασμός συγγνώμη, μεταξύ του ΟΗΕ και της πολύ περιορισμένης ομάδας του G20 θα έπρεπε να είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος, τουλάχιστον για να αντιμετωπίσουμε σε μια πρώτη γενική ε, φάση αυτό το θέμα και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Τι συμβαίνει όμως. Το G20 δεν έχει εξοπλιστεί με μόνιμες δομές γραμματείας, ε, οργάνωσης ε, και διαχείρισης των προβλημάτων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε οριστικές λύσεις. Παραμένει λοιπόν πάντα σε μία κατάσταση προαποφάσεων και επομένως και εξαιρετική δυσκολία. Πρέπει να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να επιλύσουμε τα προβλήματα είναι ο ΠΟΕ. Είναι ο χώρο στον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Επομένως δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχουμε μια έδρα συζήτησης, διότι ο ΠΟΕ είναι όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε εκπροσώπους από όλες τις πλευρές. Ακούμε και τη φωνή των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και των ισχυρών χωρών. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Επομένως δεν μπορώ ειλικρινά να σας πω ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα επί του θέματος. Και αυτή είναι η απάντηση και στον κύριο Ταραμπέλα που έθεσε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Δαντά μας είπε «Μα δεν το είχαμε προβλέψει ότι θα έρθουν η Κίνα και η Ινδία». Ναι, ναι, το είχαμε προβλέψει, αλλά νομίζαμε ότι θα ήταν πιο ελαστική η προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε φανταστεί, δεν είχαμε διανοηθεί ε, την ταχύτητα της απάντησης, όχι τόσο την αύξηση των εισοδημάτων τους, αλλά το γεγονός ότι θα αλλάξει ο τρόφος διατροφής μας. Το πέρασμα προς τις πρωτεΐνες μας κανένας δεν το είχε εκτιμήσει ανάλογα με το μέγεθός του και εκεί άλλαξε και η ε, πλέον ζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Ντόρφμαν, εγώ θεωρώ ότι ένα μεγάλο τμήμα της εγκατάλειψης της γης είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Εγώ μελετώντας τα θέματα αυτά μπορώ να σας πω ότι το μεγαλύτερο τμήμα των εκτάσεων καλλιεργήθηκε κατά το μεγάλο λοιμό το 1800. Ε, πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες ήταν κτηνοτροφικές σε μεγάλο βαθμό και ε, ήταν δάση και βουνά και το να επανέλθουμε πλέον στα δάση και στα βουνά δεν είναι το περίεργο, το παράδοξο. Το θέμα όμως τι γίνεται. Όταν πηγαίνουμε στο καύσιμο, όταν περνάμε πλέον στο καύσιμο για εκτάσεις οι οποίες είναι απολύτως παραγωγικές και γόνιμες. Δεν μπορεί να ε, φανταστούμε ότι θα ζητούμε από τους ε, γεωργούς να καλλιεργήσουν ε, ένα άγωνο τμήμα ε, ενός βουνού μιας ορεινής έκτασης, αλλά θα, γιατί θα ξαναγυρίσουμε στην συζήτηση που κάνουμε πριν. Δεν μπορεί να είναι προσοδοφόρα η καλλιέργεια μιας τέτοιας έκτασης που είναι περιθωριακή. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με την ερώτηση που έγινε για τη χρήση, ε, τη σωστή χρήση των, ε, για την εξυγίανση των εκτάσεων που έκανε ο κύριος Πρόντι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος ε, για την κοινωνία και θα πρέπει να σκεφτούμε σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο τη γεωργική χρήση αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει καθαρισμός ε, αυτών των εκτάσεων και για λόγους περιβαλλοντικής υγείας. Και ιδίω διότι εμείς κατευθυνόμαστε προς ανάπτυξη των πόλεων, αστική ανάπτυξη, η οποία είναι πλήρως ασύμβατη με αυτό που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή. Η αστική χρήση αυξάνεται και επειδή ε, η ανθρωπότητα στα δύο τρίτα της αζή της πόλης στα μέσα του αιώνα θα έχουμε ε, μια περαιτέρω έκταση πόλεων την οποία απολύτως θα πρέπει να προβλέψουμε και να φροντίσουμε να διατρέφεται. Βέβαια ο κύριος Μποβέ πολύ σωστά έλεγε ότι το θέμα της παραγωγικότητας αφορά περισσότερο και τις φτωχότερες χώρες και, τις, ε, και όχι τόσο τις πλουσιότερες χώρες. Αλλά υπάρχει και θέμα παραγωγικότητας και για τις πλούσιες χώρες που δεν έχει σχέση με τις γενετικό τροποποιημένους οργανισμούς ή με οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με τη χρήση της γης, ε, με το θέμα της υγείας των ζώων, με τους σπόρους και την τεχνική πρόοδο που είχε κάποιες πολύ ε, σημαντικές εχμές ε, ανάπτυξης τη δεκαετία του 60 και του 70, μετά είχαμε μια στασιμότητα και πλέον έχει μειωθεί η ένταση της έρευνας για τη γεωργία. Είναι πολύ λογικό λοιπόν ότι αφορά τις φτωχότερες χώρες και πρέπει να δώσουμε και την δέουσα προσοχή στην διάδοση των καινοτομιών, αλλά οι καινοτομίες αφορούν και τις ε, πολύ αναπτυγμένες χώρες. Το θέμα της ε, διατροφικής κυριαρχίας των χωρών. Eh, Αυτό ε, έρχεται σε αντούκριση, σε αντίφαση με την παραγωγικότητα. Ας δούμε την ακτή του ελεφαντοστούν, για παράδειγμα. Πρόκειται για πολιτικό δικαίωμα, λέει ο κύριος Μποβέ εκτός ε, μικροφόνου. Εντάξει, λέει ο κύριος Πρόντι, είναι σοβαρό. Δεν είναι μόνο ε, πολιτικό, είναι η συλλογική απάντηση στο ατομικό δικαίωμα, στο ανθρώπινο δικαίωμα. Νομίζω ότι από αυτού δεν μπορώ να έχω καμία ένσταση. Το θέμα τώρα που έθιξαν ο κύριος Νικολέσκου και ο Πολωνός Ευρωβουλευτής που αφορά κυρίως τις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τάση να ε, είναι ισότιμα τα κίνητρα είναι αναπόφευκτο διότι είναι θέμα δικαιοσύνης. Ξέρω ότι στις εργασίες σας υπάρχει μία τάση να ε, φτάσουμε σε ισότιμο επίπεδο και αυτό απαντά και μερικώς. αλλά απαντά και στα όσα έλεγε ο κύριος Νικολέσκου. Δηλαδή ότι όταν υπάρξει αυτή η ισορροπία, σαφώς θα υπάρχει και περισσότερο οικονομικό ενδιαφέρον για πιο ισχυρή γεωργία και σε χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβενία, χώρες οι οποίες ε, ε, εσείς αναφέρετε ως χώρες που κινδυνεύουν. Μην ξεχνάμε ότι αυτά περνάνε. Και μία τελευταία ερώτηση που μου έκανε ο κύριος ε, Δεσιλβέστρης Αυτά όλα ε, λύνονται με μια πολιτική που θα επικεντρώνεται στους νέους. Ο πληθυσμός γυράσκει, η γύραση της κοινωνίας ε, συνεχίζεται και ε, το μόνο που μπορούμε να έχουμε είναι μια σύγχρονη γεωργία. Και φυσικά η τεχνολογία και η καινοτομία εφαρμόζεται μόνο από νέους γεωργούς και αυτό κατ' εμέ περνάει από συγκεκριμένα κίνητρα, από την οικογένεια, από την επομόρφωση της οικογένειας και είναι κίνητρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την τιμή του αγαθού, αλλά είναι κίνητρα τα οποία είναι συγκεκριμένα για να μπορέσουν να ενταχθούν και νέες κατηγορίες στη γεωργία. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εισαγωγή στη γεωργία άλλων ανθρώπων που ασκούν άλλα επαγγέλματα, που σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν είναι τόσο ε, συχνά, αλλά ακόμα και η επιστροφή στη γεωργία πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κίνητρα, διότι ε, πολλές φορές ε, ε, η γεωργία απαιτεί και υψηλό επίπεδο μόρφωσης και προετοιμασίας. Κάποιος με ρώτησε αν θα επαναλάμβανα τις ίδιες θέσεις αν ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε όλη αυτή η συζήτηση είναι εκτός πραγματικότητας. Ε, η αύξηση του προϋπολογισμού και το γεγονός ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ισχυρή ενώπιον της ανάγκης να εξισορροπήσουμε τα πράγματα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ε, από οικονομικής πλευράς οι διάφορες χώρες είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτω πάντα στον εαυτό μου, πρέπει να θέτουμε όλοι και πρέπει να το θέτουμε και για το μέλλον. Ο προπολογισμό της Καλιφόρνια δεν είναι καλύτερος από τον προπολογισμό της Ελλάδος. Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένη στην πολιτική μας ανάλυση. Αλλά είναι διαφορετικό το σύστημα και δίνει μια διαφορετική ισχύ και διαφορετική δυνατότητα διαλόγου στον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της πολιτικής ισχύω της Ευρώπης και τα θέματα του προπολογισμού και όχι μόνο η αλλαγή της διακυβέρνησης την οποία θα πρέπει να θέσουν ως ερώτημα οι μελλοντικέ γενίες διότι αλλιώς εμείς πραγματικά θα εξαφανιστούμε από προσώπου γης και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις ανά τον κόσμο. Ήταν και λίγο προκλητική ερώτηση. Μου την έθεσε και ένας Κινέζος φοιτητής όταν εξηγούσα την ε, εξέλιξη του ευρωπαϊκού είδου με διέκοψε ο Κινέζο αυτό φοιτητή και μου είπε «Κύριε καθηγητά, για εξηγήστε μου καλά, η Ευρώπη τι είναι, εργαστήριο ή μουσείο» Όταν μου τέθηκε αυτό το ερώτημα, στο British School της Σανγκάη, πραγματικά προβληματίστηκα, διότι αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που μας αντιλαμβάνονται προς τα έξω είναι ότι είμαστε ένας κουρασμένος μηχανισμός, έχουμε το λαμπρό παρελθόν, είμαστε το εργαστήριο των νέων πολιτικών του κόσμου, προωθήσαμε πράγματα, αρχίσανε να αλλάζουν οι έννοιες, το καθεστώς της βετσφαλίας, όλα αυτά λίγο-λίγο και ξαφνικά πρέπει να προσέξουμε γιατί γινόμαστε μνημείο, μουσείο. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο συνειδητοποιημένοι και να έχουμε και λίγο γνώση του τι εικόνα δίνουμε προς τα έξω. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάποιες προσπάθειες πολύ πιο ισχυρές, να ενθαρρύνουμε και τις διαπραγματεύσεις της Δόχα, διότι είναι ο χώρος στον οποίο εκπροσωπούνται όλες οι χώρες και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στον οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Τέλος. Αναφέρθηκε το θέμα της έρευνας και αναρωτηθήκαμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν και δημόσιες παρεμβάσεις στην έρευνα. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν. Κάποιοι τομείς έρευνας είναι τόσο καινοτόμοι που όπως για παράδειγμα στη βιολογία και στην ιατρική, η δημόσια δέσμευση σίγουρα θα πρέπει να συνοδεύει και την ιδιωτική δέσμευση. Υπάρχει και το θέμα του land grabbing, της αρπαγής της γης, το οποίο, το επαναλαμβάνω, είναι πολιτική ανάγκη κάποιων χωρών για να διασφαλίσουν το διατροφικό μέλο των πολιτών τους. Πρόκειται λοιπόν για μία τάση την οποία εάν δεν φροντίσουμε να βάλουμε μία τάξη στην αγορά παγκοσμίω, θα δούμε να αναπτύσσεται δυστυχώς περαιτέρω στο μέλλον. Σημειώνω και συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις που έγιναν για το θέμα της κατασπατάλησης. Διότι θεωρώ ότι αυτό το ποσοστό του 20% που ε, αναφέρεται είναι ίσως αυτή τη στιγμή... Ε, υποτιμημένοι και είμαστε πολύ πάνω από το 20%. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να το επαληθεύσουμε το στοιχείο αυτό και αν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πετάμε θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ε, οικονομία. Τέθηκε και το θέμα των επιδοτήσεων και των ε, ε, πρημοδοτήσεων των εξαγωγών και τη σχετική αύξηση τιμών. Θεωρώ ότι το να ε, παίζουμε με τους περιορισμούς και τις ε, ενισχύσεις της εξαγωγές ε, δημιουργεί πολύ πιο ισχυρά φαινόμενα στρέβλωσης και όχι μόνο δεν αντισταθμίζουν αλλά δημιουργούν και πιο ισχυρά προβλήματα για τις στρεβλώσεις αυτές. Για το περιβάλλον τώρα και πάλι η συζήτηση είναι η ίδια. Πρόκειται για δημόσια αγαθά και πρέπει να την χάνουν ειδική μεταχείριση. Δεν μπορούμε να δώσουμε στη γεωργία το βάρος να υποστηρίξει αυτό το κόστος το οποίο είναι δημόσιο και σε πολύ μεγάλα μέρη του κόσμου έχουν σημαντική βαρύτητα. Η απερίμωση που αναφέρθηκε εδώ είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα της υποσαχάριας Αφρικής διότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και κάποιες ταχύτητες τις οποίες δεν θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να δούμε στο παρελθόν. Αυτά λοιπόν ως απάντηση γνωρίζω πολύ καλά ότι θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι Έχουμε περιορισμένο προπολογισμό, επομένως είναι αδύνατον, όπως είπε ο κύριος Βολέσκι στην παρέμβασή του, να κάνουμε μεγάλες πρόοδους, αλλά από την άλλη έχουμε πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους μας. Εν κατακλείδη μια παρατήρηση. Και εδώ αντλώ το παράδειγμα από τους πολύ δύσκολες διαπραγματεύσει στην Τόχα. Η Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου, επειδή εκφύσεων είναι το εργαστήριο του κόσμου, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι μία ολοένα και ισχυρότερη εντολή, μία πολύ πιο ισχυρή δέσμευση της Ευρώπης να είναι ο διαμεσολαβητής αλλά και με συγκεκριμένε θυσίε, οι οποίες όμως είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχουμε ειρήνη και ισορροπία μακροπρόθεσμα είναι πολύ σημαντική. Χωρίς αυτή τη διαμεσολάβηση το land grabbing, οι ενισχύσεις, οι απρόβλεπτες για τις εισαγωγές ή και το γεγονός των επιδοτήσεων σε περίπτωση κρίσης θα γίνουν αναποφευκτές. Για αυτές λοιπόν τις τόσο επιζήμιες και σημαντικές πτυχές μπορούμε να βρούμε λύση μόνο εάν καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η ευρωπαϊκή συνεισφορά για τη συμφωνία αυτή, κατά την άποψή μου, είναι ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόντι, ευχαριστούμε όλους και υπενθυμίζω στις 2 ξεκινούν οι ψηφοφορίες. Πέρα συνεδρίαση.